Καλημέρα σε όλους. Έπρεπε να περιμένω λίγο να έρθουν κάποιοι συνάδελφοι για να αρχίσουμε. Θα ήθελα να σας ενημερώσω όλους τους συναδέλφους και τους συμμετέχοντες ότι θα ε, έχουμε απευθείας μετάδοση από το διαδίκτυο και ήχου και εικόνας. Πρέπει πρέπει να σας ρωτήσω αν ε, δέχεστε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Μάλιστα, το σχέδιο λοιπόν έχει διανεμηθεί στις 21 Μαΐου. Κατόπιν ετοίματος των συνσηγητών Φόξ και Χέφνερ προτείνω αύριο στο τέλος του πρωινού να συζητήσουμε το θέμα που αφορά ε, τις έδρες των ε, θεσμικών οργάνων. Ε, έχετε λάβει όλη αυτή την ειδοποίηση και παρακαλώ να τη δεχτείτε. Ο καθορισμός της έδρας των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το θέμα για αύριο. 11.30 με 12.30. Και θα σας πρότεινα λοιπόν αμέσως μετά τη συζήτηση του θέματος του κυρίου Κασίνη να συζητήσουμε αυτό το θέμα ο καθορισμός της έδρας των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνείτε. Κύριε ε, ε, Χέφνερ, για το δικό σας θέμα ε, κάνω ανακοίνωση για να δούμε αν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για να αλλάξουμε έτσι την ημερήσια διάταξη. Επαναλαμβάνω, για να βεβαιωθούμε ότι το καταλάβαμε όλοι, 11.30 με 12.30 αύριο το πρωί μπορείτε. Α, νωρίτερα, 10 και μισή, 10 και 35 μάλιστα. Συμφωνείτε. Ο κύριος Χέφνερ, εμείς το είχαμε ζητήσει από την πρώτη μέρα πριν από ένα μήνα και πλέον. Ε, υπήρξε κάποιο πρόβλημα, ένα σπάλμα επικοινωνίας στη γραμματεία, γι' αυτό και πάλι έπρεπε να αλλάξει. Έχει προαποφασιστεί αυτό, θα πρέπει και πάλι να το αλλάξουμε. So then you agree with my suggestion that... Άρα συμφωνείτε με αυτό που προτείνω εγώ, μάλιστα. Λοιπόν, οι υπόλοιποι συμφωνούμε. Καλώς. Λοιπόν. Okay. Okay, that's fine. So, uh, as we got a very proper request... Λοιπόν, έχουμε αυτό το αίτημα των δύο εισηγητών για τον καθορισμό της έδρας των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανονικά έπρεπε να συζητηθεί αύριο 11.30 με 12.30. Δεν τους βολεύει, διότι έχουν και άλλη έκθεση αλλού. Γι' αυτό θα το εξηγήσουμε μία πρόταση. Ποια ήταν ε, η πρόθεση και έχετε το πρόγραμμα και μάλιστα γραπτό ε, που συζητούν πάντα οι συντονιστές με τη γραμματεία να γίνει σήμερα η ακρόαση και αύριο υπό το φως της ακρόασης να γίνει συζήτηση μεταξύ μας. Έτσι, δεν ήταν, έτσι είχαμε συνεννοηθεί και ε, η γραμματεία μπερδεύτηκε, το έβαλε αντίστροφα και παρακαλούμε να διορθωθεί όπως το είχαμε αποφασίσει. Σήμερα ακρόαση, αύριο συζήτηση. Έτσι έχει τώρα η πρόταση και συμφωνούμε όλοι σήμερα η ακρόαση, αύριο συζήτηση, λέει και ο κύριος Γκουαλτιέρη. Μάλιστα. Για να το διευκρινίσουμε. Ο κύριος Φόξ μας είπε ότι αύριο στις 11.30 κολλείεται. Γι' αυτό μας ζήτησε. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Ότι μας ήρθε και ένα νέο αίτημα. Και ακριβώς επειδή είναι τόσο σημαντικό το ζήτημα, προτείνω ε, να προταχθεί αυτό. Και εγώ σας συνιστώ γιατί θεωρώ ότι είναι το θέμα πάρα πολύ ε, ευαίσθητο, να συμφωνήσουμε ότι αμέσως μετά ε, τις ανακοινώσεις σχετικά με τις τάσεις των ε, συντονιστών να έχουμε αυτό το πρώτο θέμα στη μερίσια διάταξη. Να είναι το 12. Μετά το 11 να γίνει 12 αυτό το θέμα, το πρώην 6. Λοιπόν, σήμερα κρόαση, αύριο Yes, yes. So my Λοιπόν, αυτή είναι η σύστασή μου και θα σας παρακαλούσα να συμφωνήσετε όλοι. Εντάξει. Και ο Ράφαλ Τσαρκόφσκι συμφωνεί. Εντάξει. Εγκρίνεται λοιπόν. Αν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Ωραία. Προχωρούμε. Το δεύτερο θέμα ανακοινώσει. Οι πολιτικές ομάδες όρισαν τους εξής ε, εισηγητές για τα θέματα που ανατέθηκαν την περασμένη συνεδρίαση. Γνωμοδότηση για πρόταση κανονισμού ε, που διέπει τη λειτουργία της Europol. Η κυρία Τέιν των Φιλελευθέρων και γνωμοδότηση ε, για την Επιτροπή Προπολογισμών για την έκθεση για τον προγραμματισμό είναι ο κύριος Μπροκ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αν δεν υπάρχουν σχόλια, θεωρώ ότι εγκρίνονται αυτοί οι διορισμοί από την Επιτροπή μας. Για να με συμφωνείτε με την πρόταση των συντονιστών. Ωραία. Ούτως και αποφασίζεται. Πώς έχει η διαδικασία κύρωσης. Ως συνήθως στο σημείο 2, στο φάκελό σας θα βρείτε ενημέρωση του εγγράφου που προετοίμασε ε, το Τμήμα Πολιτικής και ευχαριστούμε πολύ ε, που αναφέρει ε, πώς έχει διαδικασία κύρωση σε κάθε κράτο μέλος για τις συνθήκες για την οικονομική διακυβέρνηση, καθώς επίσης και τη συνθήκη για την προσχώρηση της Κροατίας. Αυτές είναι οι ανακοινώσεις. Σε ό,τι αφορά το τρίτο τμήμα, το τρίτο σημείο μάλλον έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων, θα ήθελα να σας πω ότι τα πρακτικά της 14ης Μαρτίου 2013 και της 18ης και 19ης Μαρτίου 2013 ε, έχουν διανεμηθεί και όσοι ήθιστε αν δεν διατυπώσετε καμία αντίρρηση μέχρι το τέλος της συνεδρίασης θα θεωρηθούν εγκριθέντα τα πρακτικά. Αν έχετε τίποτα να πείτε να μας το πείτε και ελπίζω πραγματικά τώρα να είμαστε σε θέση να μπούμε στο σημείο 4, παρουσία του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χαίρομαι που σας βλέπω πάρα πολύ. Στις 16 Μαΐου η διάσκεψη των Προέδρων ενέκρινε ε, την έκθεση DAF ε, υπομορφή νομοθετικής πρωτοβουλίας σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 48 του κανονισμού μας. Αυτή η αλλαγή είναι διαδικαστική και δεν απαιτεί καμία σημαντική τροποποίηση των εγγράφων που ενδεχομένως να είχαν εμποθήσει να γίνει αύριο όπως είχε προβλεφθεί η ε, ψηφοφορία. 79 τροπολογίες έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα από τους Ρανζέλ Γκουρμάη, Γκούσταυσον, Μέσερ, Σμιτ, Λαμασούρ, Λεγκρίπ, Σόπλ, Σόλτς, Κασίνη, Γιαννάκου, Λάινεν, Μορέρα, Χιόρκμαρκ, Τσασκόφσκι, Κάρας, Ζέμπερ, Χέφνερ, Βίλαντ, Οντί και από τον ίδιο τον εισηγητή τον κύριο Νταφ. Υπό την έννοια αυτή, οφείλω να σας υπενθυμίσω ότι η διάσκεψη των Προέδρων επέμεινε ότι η έκθεση δεν θα πρέπει να υπερβεί ε, το πεδίο που ορίζεται στον τίτλο που είναι η δημοκρατική και αποτελεσματική διεξαγωγή των ε, εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διότι στην πραγματικότητα ορισμένε από τι τροπολογίε που κατατέθησαν φαίνεται να υπερβαίνουν αυτό το πλαίσιο και έχουν να κάνουν με πολιτικέ διαβουλεύσει κατόπιν των εκλογών. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Ντάφ, για να μας παρουσιάσει τη θέση του ε, ε, επί των τροπολογιών και ενδεχομένως να μας ε, πει και ποιες προτάσεις έχει για συμβαστικές τροπολογίες. Παρακαλώ, με μεγάλη χαρά σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Um, Καλησπέρα σε όλες και όλους σχετικά με τα ανακοινοθέντα της διασκέψης των Προέδρων μου φαίνονται λαβυρινθώδη. Δεν νομίζω ότι κατενόησαν καν την φύση του εγχειρήματος που έχει αναλάβει η Επιτροπή Συνταγματικών. Η διάσκεψη των Προέδρων αναχέτησε έτσι νομοθετική έκθεση για την εκλογική διαδικασία του Κοινοβουλίου παρόλο που αυτή ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία στην Επιτροπή Συνταγματικών. Με κάθε σεβασμό βεβαίω, εγώ θα συνεχίσω και θα περιγράψω τα όσα θεωρώ ότι έχουμε στο σχέδιο που είναι σαφώς βελτιωμένα με τις 85 τροπολογίες. Έξι από την κυρία Μπελιέ. που κατατέθηκαν μετά την λήξη της ημερομηνία. Ωστόσο θα παρακαλέσω την Επιτροπή Συνταγματικών να τις δεχθεί. Να ψηφιστούν δηλαδή. Αν και το θέμα αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε αύριο το πρωί. Έτσι λοιπόν θυμίζω ότι πρόκειται για πολιτικού χαρακτήρα ψήφισμα μετά από απόφαση Συμβουλίου και Κοινοβουλίου να προτάξουν την ημερομηνία, καθώς επίσης και την απόφαση του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν να ενθαρρύνουν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να προβούν σε προβολή υποψηφιωτήτων για την Προεδρία της Κομισιόν στα πλαίσια της προεκλογικής τους εκστρατείας. Το δε κοινοβούλιο το δέχθηκε αυτό με σημαντική πλειοψηφία ήδη το φθινόπωρο. Και αυτό που απαιτείται τώρα είναι να κατανοήσουμε ορισμένες από τις πρακτικές επιπτώσεις της αποφάσεως αυτής. που συνδέονται με την οργάνωση της προεκλογικής εκστρατείας επειδή θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της εκστρατείας ώστε να τονιστεί η ευρωπαϊκή διάσταση, να βελτιωθεί η διαφάνεια και να ενισχυθεί η συμμετοχή του εκλογικού σώματος στην εκλογή. Γι' αυτό θέλουμε αυτές τις υποψηφιότητες για Προεδρία της Κομισιόν που να προταθούν από πλευράς των, των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δράσει με τρόπο ευφυή και γρήγορο, καθώς και θαραλέο, για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τις νέες εξουσίες που του προσφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας. Έτσι ώστε να διαμορφώσει την Επιτροπή σε πρώτο βαθμό ιδίως εκλέγοντας διάδοχο του Πρόεδρου Μπαρόσο ήδη από τον επόμενο Ιούλιο, ώστε να συμμορφωθούμε έτσι και με το χρονοδιάγραμμα της συνθήκης, το οποίο προβλέπει η Κομισιόν έχει ήδη αναλάβει από 1η Νοεμβρίου. Σήμερα, όπως κάναμε και το 2009, μπορούμε να αναβάλουμε την εκλογή του Πρόεδρου της Κομισιόν μέχρι τον Σεπτέμβρη. Αυτό θα είναι μεγάλο λάθος όμως, διότι δεν θα έχουμε συγκροτημένη σε σώμα επιτροπή, Κομισιόν δηλαδή, μέχρι τον Νοέμβριο. Και σε καιρούς έντονης οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής δυσχέρειας που σημειώνεται στην Ένωση, Χρειαζόμαστε κομισιόν και μάλιστα ισχυρή κομισιόν και όσο δυνατόν συντομότερα. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν να διεξέλθω εν συντομία τις συμβαστικές τροπολογίες καθώς και ορισμένες από τις πιο σημαντικές και πρώτα θα σας ευχαριστήσω για, τη συνεργασία που ήταν πραγματικά πρώτη τάξης. Έχω διανύμει την λίστα ψυχοφορίας. Έχω την 3 έπειτα της παραγράφου 1 πρώτα που αναφέρεται στον χρόνο πρώτων εκλογών όπου θα χρειαστεί να είναι ήδη δημόσια γνωστές οι υποψηφιότητες. Αυτό το θέμα είναι περίπλοκο και ένα είδος λαχείο. Διότι ο συμβασμός που πρότεινα ή που προτείνω είναι να είναι δημοσιευμένες οι υποψηφιότητες, δηλαδή τα κόμματα να έχουν δημοσιεύσει τα ονόματα των υποψηφίων τους 8 εβδομάδες πριν από την ψηφοφορία. Επισήμως τώρα σε ορισμένες χώρες δεν είναι αναγκαίο να δημοσιευτούν τα ονόματα αυτά τόσο νωρίς. Στην Ιταλία νομίζω υπάρχει και νόμος που λέει πέντε εβδομάδες. Τονίζω ωστόσο ότι αυτό αφορά την επίσημη δημοσιοποίηση από πλευρά Ιταλικού κράτου. Ενώ εδώ μιλούμε εμεί για τα πολιτικά κόμματα. ώστε αυτά να κινηθούν διαφανώς και με ταχύτητα για την επιλογή και δημοσίευση των υποψηφιωτήτων. Ίσως μπορούμε να βελτιώσουμε τη διατύπωση έτσι ώστε να φανεί καθαρά ότι απευθυνόμαστε πρωτίστως στα πολιτικά κόμματα. Γυρνώντας σελίδα, συμβαστική 4, εδώ δέχομαι την ιδέα αυτή της κυρία Σέπφλιν ώστε όσοι κατέρχονται ως υποψήφοι να αναλάβουν τις εντολές τους εφόσον εκλεγούν διότι στο παρελθόν υπήρξαν πολλά μεγάλα ονόματα κομμάτων που μπήκαν πρώτοι στις λίστες χωρίς να διαθέτουν απολύτως καμία πρόθεση να καταλάβουν έδρα στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό ίσως ήταν κάτι που μπορούσε να το κάνει δεχτό κανείς σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προ ετών. Αλλά τώρα αυτό θα σήμαινε μια κίνηση εξαπάτηση του εκλογικού κοινού. Ο ψηφοφόρο είναι απαραίτητο να μπορεί να δει ποιον θα βάλει σε έδρα στο κοινοβούλιο. Ερχόμαστε μετά στην ισορροπία των φύλων στους καταλόγους υποψηφίων. Εδώ είχα πολλές τροπολογίες προς την αυτή κατεύθυνση. Και από εσά την ίδια κυρία Πρόεδρε, η κυρία Προεδρεύουσα, από την Σαντρίν, και από άλλους, Λαμασούρ και Λεκρύπ. Εγώ θεωρώ ότι η τροπολογία 40 Λαμασούρ και Λεγκρίπ όντως ποιείται χρήση της σωστής ορολογίας και αποπνέει το σωστό πνεύμα. Δεν μπορούμε να βάλουμε εκλογικές ποσοστώσεις στις χώρες μέλη. Ίσως θα έπρεπε, αλλά δεν μπορούμε. Είπα από την αρχή ότι δεν πάμε να αναδιατυπώσουμε το εκλογικό δίκαιο της Ένωσης. Στρέφουμε απλώς τα πολιτικά κόμματα και τις χώρες μέλη στην κατεύθυνση που επιθυμούμε αυτά να ακολουθήσουν. Ωστόσο μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό. Εγώ πάντως γενικά δέχομαι την ιδέα Να προσπαθήσουμε δηλαδή να επιτύχουμε καλύτερη ισορροπία φύλων. Αυτό θα σημάνει για ορισμένου ισότητα. Στη δική μου αντιπροσωπεία οι άνδρες βρισκόμαστε στην μειοψηφία και ξέρω πολύ καλά γιατί σα μιλώ. Συμβαστική τώρα 5 αφορά το μορφότυπο του ψηφοδελτίου. Και αυτό περίεργο είναι περίπλοκο θέμα, διότι σε ορισμένες χώρες μέλη αυτό το φόρμα, ο μορφότυπος, το σχέδιο είναι ζήτημα πρωτογενούς δικαίου. και θα είναι επομένως αδύνατο για τις χώρες αυτές να μπορέσουν να συμφωνήσουν με την πρότασή μας ώστε τα ονόματα και σύμβολα των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων εμφανίζονται στα ψηφοδέλτια αυτά. Και εδώ πάντως υποδεικνύουμε μια κατεύθυνση που επιθυμούμε να ε, λάβουν τα κόμματα. Θα είναι δε ενδιαφέρουσα δοκιμασία για τις σχέσεις μεταξύ των ομοσπονδιακών πολιτικών κομμάτων στο ευρωπαϊκό επίπεδο και των συνδεδεμένων κομμάτων μελών στο εθνικό επίπεδο να ειδούν δηλαδή εάν θα καταφέρουν να συμφωνήσουν πάνω σε μια κοινή εκστρατεία. Συνεχίζω. Συμβαστική 6 την οποία εμπνεύστηκα από τέσσερις καλές τροπολογίες που μιλούν για την αναγκαιότητα να γίνει εκστρατεία πάνω σε κομματικές πλατφόρμες για τους υποψηφίους δηλαδή και την Προεδρία της Κομισιόν. Θα έχουν αυτοί βέβαια και δικό τους πρόγραμμα, δεν αμφιβάλλω, αλλά θα συμφωνήσουν ωστόσο ε, να σταθούν και να κινηθούν πάνω στις ευρύτερες εκλογικές πλατφόρμες των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Για την παράγραφο τώρα 3α νέο, εδώ υπάρχουν οι τροπολογίες 48, 47 και 50 του Τζέραλτ είναι η ευρύτερη του Γκέραλτ Χέφνερ που μυστική ψηφοφορία μέσα στα ίδια τα κόμματα για την εκλογή του υποψηφίου για την Προεδρία της Κομισιόν. Έχω κατανόηση για την ιδέα αυτή. Βρίσκω όμως ότι είναι κάπως πρόορη. Ας είμαστε ρεαλιστές, όσο και φιλόδοξοι, και ας πειραματιστούμε πρώτα. Να δούμε εάν θα μπορέσουν έτσι να χειριστούν τα της δημοκρατίας. Είναι ένα πρώτο πείραμα για την επιλογή και πρόθεση αυτών των υποψηφιωτήτων. Θα είναι μια λεπτή και βέστη διαδικασία. Ελπίζω να είναι δημοκρατική και ελπίζω να είναι και διαφανής. Είδα ότι οι πράσινοι θα κάνουν προκριματικές εκλογές. Αυτό είναι συναρπαστικός ιδέα και σας εύχομαι καλή τύχη. Αλλά δεν απαραίτητα και το ορθότερο για όλα τα πολιτικά κόμματα. Με την άδειά σας προτιμώ τη δική μου 47. Τώρα για τις εκπομπές σχετικά με τις εκλογές. Εδώ είχαμε πέντε τροπολογίες. Συν μία πρόταση του κ. Μέσσερ Σμιτ να διαγραφεί ολόκληρη παράγραφος. Ξέτασα βέβαια όλες τις τροπολογίες προσεκτικά. Αλλά παρόλα αυτά προτιμώ τη δική μου αρχική διατύπωση δηλαδή οι χώρες και τα κόμματα να επιτρέψουν στους δημόσιους φορείς να μεταδίδουν τα κομματικά πολιτικά μηνύματα στην διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Η συμβαστική 7 είναι αρκετά καθαρή. με την έννοια ότι η σύνταξη των ψηφοδελτίων θα πρέπει να βρει τα κόμματα ενεργά, proactive δηλαδή, να βρουν πολίτες Ευρωπαίους πολίτες που να κατοικούν σε χώρες άλλες εκτός της δικής τους για να τους περιλάβουν ως υποψηφίους στις λίστες τους. Κάτι τέτοιο θα βελτιώσει πολύ τον υπερεθνικό χαρακτήρα της εκλογής. Και αν επιμένουμε οι χώρες μέλη να σεβαστούν τον νόμο που είναι ξεκάθαρος εν προκειμένου. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε και τα πολιτικά κόμματα να εμφυσίσουν ζωή στην ιδέα αυτή. Ε, κυρία Γκουρμάη, αν μπορείς να επιταχύνεις Άντζου σε παρακαλώ, διότι έχω πολλούς που αδειμονούν να λάβουν το λόγο και βέβαια είναι σημαντικό να ακούσει όλα τα σχόλια. Κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ, αλλά πρέπει να σα εξηγήσω περί τίνο πρόκειται. Η 8η αναφέρεται στην ημερομηνία των εκλογών, της ε, εκλογής δηλαδή. Η τροπολογία 69 καθορίζει το πιθανό χρονοδιάγραμμα για όσα θα χρειαστεί να γίνουν Ιούνιο και Ιούλιο, έκτο και έβδομο μήνα. Βεβαίως δεν θα γίνει τίποτε το επίσημο πριν από την συγκρότηση σε σώμα του νέου κοινοβουλίου. Αυτό είναι απόλυτα θεμελιώδες και οφείλουμε να το τονίσουμε, διότι αν δεν το πράξουμε τότε θα μας τσαλαπατήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Νομίζω ότι σε αυτά που είπα περιέλαβα όλες τις πιο σημαντικές, ας πούμε όλες είναι σημαντικές, αλλά τις πιο θεμελιώδεις τροπολογίες. Και συμβαστικές και απλές. Θα σταματήσω λοιπόν εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, είδα ότι όλα είναι και περισσότεροι συνάδελφοι θέλουν να σχολιάσουν και φυσικά και θέλουμε να ακούσουμε και την ε, περίληψη που θα κάνει στο τέλος. Ο Ρομπέρτο είναι ο πρώτος που παίρνει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ομάδα μας ε, καλωσορίζει τις συμβιβαστικές και εν γέννη είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα της συζήτησης. Ανάμεσα στους ε, σκιώδεις και στον ε, εισηγήτη, αλλά έχω κάποιες παρατηρήσεις που θα ήθελα να σας αναφέρω. Η πρώτη είναι βεβαίως αυτή που ανέφερε και ο Άντριου και αφορά το θέμα των εκτός θέματος ε, τροπολογιών. Εκτός θέματος ε, όσον αφορά το πεδίο που ορίζει ο τίτλος. Νομίζω θα πρέπει να σημειώσουμε το γεγονός ότι η διάσκεψη των Προέδρων μας ζητά να ακολουθήσουμε πιστά την εντολή και εν γέννη πρέπει να πω ότι δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα για να εγκαταλείψουμε αυτές τις ε, τροπολογίες. Πιστεύω πως υπάρχει το θέμα της τροπολογίας 69 ε, που μπορεί όμως να λυθεί μόνο με έναν τρόπο. Γιατί διαφορετικά είτε δεν θα ψηφιστεί, δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία ή αν τεθεί σε ψηφοφορία η ομάδα μας θα καταψηφίσει. αφορά τη δέσμευση του Κοινοβουλίου για έναρξη διαπραγματεύσεων περί της δήλωσης 11, ε, αλλά χωρίς να γίνεται καμιά δήλωση για το περιεχόμενο. Αυτό είναι το μάξιμο που θα μπορούσαμε να δεχτούμε και θα ήταν σοφό να το κάνουμε αυτό, γιατί διαφορετικά ούτως ή άλλως από πολιτικής άποψης αυτή η τροπολογία θα απορριφθεί. Μπορούμε να το υποβάλουμε εμείς για προφορική τροπολογία, ε, πάση περιπτώσει μπορούμε να συμφωνήσουμε μεταξύ μα. Πάντω, αυτό είναι το μάξιμο που μπορούμε να πούμε για αυτό το θέμα, που δεν αφορά πρακτικέ ρυθμίσει για τι εκλογέ, αλλά αφορά την περίοδο μετά τι εκλογέ. Ε, αυτό σημαίνει επίση ότι σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να ε, εξοικονομήσουμε τη 2 και την 26, δηλαδή το εκτιμώντα και το τις αιτιολογικές σκέψεις, ενώ βεβαίως οι 74, 73 και 77 θα πρέπει να απορριφθούν γιατί είναι γραφειοκρατικής φύσης ή διαφορετικά θα τις απορρίψουμε. Δεύτερη παρατήρηση. Αυτό το θέμα μπορεί και από πολιτικής άποψης να επιληθεί. Από τη γνώμη μου, οι τρεις τροπολογίες 71, 75 και 78 για την ενιαία ημερομηνία για τις εκλογές από τον ε, συνάδελφο Ραζέλ θα μπορούσαν ε, και επίσης να καταπέσουν μετά από την έγκριση της συμβιβαστικής Α γιατί τεχνικώς ε, μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν καλύπτεται, αλλά από πολιτικής άποψης η συμβιβαστική είναι ένας τρόπος για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα με την ενιαία ημερομηνία χωρίς να την έχουμε την ημερομηνία που φυσικά μπορεί να είναι πιθανό να μην γίνει δεκτό από τα περισσότερα κράτη-μέλη. Έχω την εντύπωση ότι ούτως ή άλλως διαφορετικά αυτές οι τροπολογίες θα απορριφθούν. Οπότε είναι αυτός ένας τρόπος να πούμε πως το πνεύμα του, της τροπολογίας του Πάολο κατά κάποιο τρόπο έχει ληφθεί θετικά υπόψη αν θεωρήσουμε πως καταπίπτει η ε, τροπολογία αυτή μετά την έγκριση της συμβαστικής. Τελευταίες δύο παρατηρήσεις που αφορούν τη συμβαστική τρία. Άντριου, ήδη εσύ πρότεινε σε μια λύση που νομίζω θα μπορούσε να σταθεί, διότι φυσικά δεν μπορούμε να φανταστούμε στην Ιταλία ούτε και στις άλλες χώρες μια αλλαγή νομοθεσίας που θα ε, θα οδηγούσε να γίνει νωρίτερα η παρουσίαση των υποψηφίων, αλλά αν κάποιο πολιτικό κόμμα επιλέξει να φτιάξει τον ε, εκλογικό του κατάλογο νωρίτερα, μπορούμε να ζητήσουμε από τα πολιτικά κόμματα να δημοσιεύσουν άμεσα τους καταλόγους, ε, τα ψηφοδέλτιά τους, και πιστεύω πως μια τέτοια αλλαγή θα ήταν καλή. Τέλος, για τη συμβιβαστική 5, εδώ και πάλι νομίζω ότι ακριβώς διότι κάποιες χώρες θα δυσκολευτούν, θα είναι περίπλοκο αν έχουμε αυτό το αποτέλεσμα μόνο μέσω τη αλλαγή τη νομοθεσία. Δεν ξέρω αν αυτό θα ήταν δυνατόν σε όλες τις χώρες, αλλά πάντως σε πολλές χώρες θα μπορούσαμε να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα με πολιτικό τρόπο μέσω απόφασης των κομμάτων να συμπεριλάβουν για παράδειγμα στο δικό του σύμβολο μια αναφορά στο σύμβολο του Ευρωπαϊκού του κόμμα, στο νέο όνομα του υποψηφίου οπότε δεν πρέπει απλά να μιλήσουμε, να απευθυνθούμε μάλλον να ασχοληθούμε με τα κράτη-μέλη αλλά και με τα εθνικά κόμματα ώστε όποτε αυτό είναι δυνατό από μόνα τους να ακολουθήσουν ε, την κατεύθυνση αυτής της τροπολογίας χωρίς να χρειαστεί νομική αλλαγή ή ένα διπλό σύμβολο ή διπλό όνομα πάνω στο ψηφοδέλτια. Αυτά είναι τα βασικά σημεία που, ήθελα, που ήθελα να αναφέρω. Κατά τα λοιπά συμφωνούμε για τις ε, συμβιβαστικές και ευχαριστούμε τον Άντριο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Σόφλιν και μετά ο Ράφαλ Τσασκόφσκι. Ευχαριστώ, ο πρόεδρε, στα Ουγγρικά, ο κύριο Σόφλιν, και συνεχίζει στα Αγγλικά. Συμφωνώ απολύτω με πολλά από όσα είπε ο Άντρου και αρκετά από όσα είπε ο Ρομπέρτο. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για την ουσία και ε, μερικά για το κείμενο. Θα θυμάται ο Άντρου ότι αυτό το έλεγε ο Ρίτσαρτ Κόρμπετ στο παρελθόν. Δεν ξέρω αν τον θυμάστε πολύ, ο Άντρου και εγώ τον θυμόμαστε. Ε, κάτι ε, που υπόθηκε και προηγουμένως. Έχει σημασία και η διαφάνεια και η συμμετοχή στις εκλογές. Εγώ θα πρότεινα να προσθεθεί και η προβολή. Γιατί και η προβολή είναι σημαντικό. Δεν είναι καθόλου εύκολο και θα πρέπει να το γνωρίζουμε. Το δεύτερο επίσης που θα ήθελα να προσθέσω είναι το σώμα των επιτρόπων θα πρέπει να έχει συγκροτηθεί πριν τις αρχές Νοεμβρίου. Μα αυτό είναι πολύ σημαντικό και την περασμένη φορά ε, είχαμε αποκλίνει λίγο για κάποιους ε, λόγους όχι και τόσο σημαντικούς. Ε, στη ουσία τώρα, αυτό που θα ήθελα να πω επίσης είναι ότι αν προσπαθούμε να κάνουμε εδώ κάτι εδώ είναι να ενθαρρύνουμε τον εξευρωπαϊσμό αυτών των εκλογών. Να καταλάβει ο κόσμος δηλαδή ότι είναι ευρωεκλογές. Δεν θα είναι εύκολο κάτι τέτοιο όμως διότι ε, βασικά εμείς πηγαίνουμε κόντρα στο ρεύμα εδώ. Τι προσπαθούμε να κάνουμε. Να καταλάβουν οι εκλογείς ότι η Ευρώπη υπάρχει. Και δεν είναι μια μεγάλη ε, γραφειοκρατία με πολλά πλοκάμια, αλλά υπάρχει και ως πολιτική δύναμη και είναι και πρωταγωνιστής ε, σε κάποια ζητήματα και θα πρέπει και οι πολίτες κάπως να συνεισφέρουν. Και δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια, πόσα χρόνια το έχουμε ξαναζήσει, δεν είναι εύκολο, θα πρέπει να δώσουμε μάχη, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία, ζωτική σημασία όσοι συμμετέχουν σε αυτές τις εκλογές να έχουν υπόψη τους και αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν επί της ουσίας. Τώρα για το κείμενο δεν είναι πολύ σημαντικά λεπτομέρειες, είναι, το έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν, για τη συμβαστική τροπολογία 3. Νομίζω με τις 8 εβδομάδες υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μου φαίνεται πολύ μεγάλο διάστημα. Το έχουμε ξανασυζητήσει, δεν ξέρουμε πώς να το ξανασκεφτούμε. Ακόμα και με τη δική σου εκδοχή που προτείνεις μόνο για τα πολιτικά κόμματα, το ζήτημα είναι πότε θα αρχίσει η συζήτηση γι' αυτό και πώς θα διεξαχθεί και δεν είμαι βέβαιος ότι είναι η σωστή περίοδο 8 εβδομάδες. Σε πάση περιπτώσει, ίσως να το ξανασκεφτούμε. Για την τροπολογία 69, συμφωνώ πάρα πολύ με τον Ρομπέρτο Γκουαλτιχέρη. Είναι κοντά του και η δική μας θέση. Στη διάσκεψη των Προέδρων ε, μπορεί να συναντήσει μεγάλη αντίσταση, μπορεί να αντιταχθούν στα νερά ε, το χρονοδιάγραμμα αυτό. Συμφωνώ πάντως με τον Γκουαλτιέρη. Και το ίδιο ισχύει ε, για την τροπολογία 73 του ΟΝΤΗ. Γιατί συμβιβαστική 7 τώρα. Η διατύπωση είναι με ευρεία και ενδεχομένω είναι εκτεθειμένη σε μια κατάσταση. Δεν να διαφωνώ, απλώ θέλω μια διευκρίνηση. Μπορεί κάποιος να είναι υποψήφιος σε μια χώρα μέλος χωρίς να έχει ε, την υπηκότητα ή την ηθαγένεια, αλλά δεν θα πρέπει να είναι κάτοικος της χώρας. Ναι, λέει ο κύριος Νταφ. Ε, δηλαδή, μπορεί κάποιος Ιρλανδός που ζει στην Πορτογαλία να κατεβεί στην Πολωνία. Μπορεί να είναι παράλογο αυτό, αλλά ο παραλογισμός έχει μια κακιά συνήθεια. Έρχεται και σε χτυπάει πισόπλατα. Ε, και Γενικά, ε, τη ε, Ράντα, Αμασούρ, Δεκρύπ και τα λοιπά, συμφωνούμε για το νέο ψηφοδέλτιο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ κύριο Τσασκόφσκι και μετά ο κύριος Χέφνερ. Πάρα πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πολύ, Άντρου. Εξαιρετική εργασία σου εδώ. Τον ίδιο στόχο έχουμε, νομίζω. You ε, θέλουμε οι ευρωεκλογέ να γίνουν και πιο ευρωπαϊκές αλλά και να έχουν σημαντικό ρόλο σε αυτό. Λοιπόν, είναι ενδιαφέρον να δούμε τι κάνουν τα εθνικά μας κόμματα, γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά όντως θα πρέπει να υπάρχει μια πάρα πολύ στεναρή θέση του Κοινοβουλίου για να επιτύχουμε όλους μας τους στόχους. Ε, Για την ε, τροπολογία 69, συμφωνώ και εγώ με τους φίλους που μίλησαν προηγουμένως. Οι στόχοι είναι σαφείς ε, και θα πρέπει να τους πετύχουμε, αλλά χωρίς ιδιαίτερη υπερέκταση όταν πρόκειται για την αντιπαράθεση στη διάσκεψη των Προέδρων. Και το θέμα με την ημερομηνία των εκλογών, γιατί τα κάνουμε όλα αυτά, για να ε, εκλεγεί όσο γίνεται πιο γρήγορα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά δεν ξέρω αν θα πρέπει να είναι τόσο αυστηρό το χρονοδιάγραμμα για τόσο δεδομένο. Μπορεί να χρειαστεί κάπως να αποφασιστεί και εκτός των πλαισίων της έκθεσης, να μην είμαστε αντιπαραγωγικοί στην προσέγγιση μας. Ένα ερώτημα, γιατί εγώ έχω κάποια αμφιβολία. Το θέμα είναι ποιος είναι υποψήφιος για τις εκλογές. Υπάρχει αυτή η ιδέα που λέγει ότι όποιος κατέρχεται σε εκλογές θα πρέπει να είναι πρόθυμος να καλύψει και την έδρα ε, εάν την κερδίσει. Το καταλαβαίνω αυτό. Ξέρω ότι υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις σε διάφορες χώρες. Ε, στη δική μου χώρα, ας πούμε, θα ήταν πραγματικά ε, θράσος κάποιος ας πούμε, να κατέβει σε εκλογές και μετά να μην εκλεγεί βουλευτής, να μην καλύψει την έδρα. Μπορεί κάποιο δηλαδή να είναι στο ψηφοδέλτιο και μετά να μεταβεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περάσει, αλλά... Αν υπάρχει λογική και αυτή ακολουθούμε ότι να μην είσαι υποψήφιο σε ένα ψηφοδέλτιο με ιστεροβουλία, δηλαδή κατεβαίνω για βουλευτή, αλλά μετά ε, θα μεταπηδήσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ή αναλαμβάνει κάποιο ένα υπουργικό θόκο. Να μην κατηγορηθεί. Δεν το έχω λύσει αυτό, απλώς σκέφτομαι φωναχτά. Κάτι που μπορεί να φαίνεται ως καλή ιδέα, μπορεί στη δική σου χώρα και τη δική μου να αποδειχθεί αντιπαραγωγικό να έρθουμε αντιμέτωποι εδώ σε μια, με μια πραγματικότητα όπου οι υποψήφοι ευρωβουλευτές στη συνέχεια γίνονται επίτροποι. Ευχαριστώ πολύ. make πολύ. Συμφωνώ με τις γενικές γραμμές της έκθεσης. Θα προτιμούσα να είναι νομοθετική η έκθεση. Είναι λίγο δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι δεν μας επιτρέπεται αυτό. Μα αν δεν μπορεί το κοινοβούλιο να λάβει εδώ την ε, πρωτοβουλία, ποιο άλλο θα το κάνει και να ορίσει και το γενικότερο πλαίσιο των ευρωεκλογών. Προσπαθεί ο εισηγητή και εμεί να κάνουμε ό,τι μπορούμε και πράγματι είναι πολύ καλή η πρότασή του. Η γενική ιδέα ποια είναι. Συμφωνούμε όλοι. Δεν θα επανέλθω σε αυτό μόνο μερικά έτσι, επιμέρους σημεία για τη συμβαστική 4. Αν μιλούμε για ψηφοδέλτιο, τον έφεραν κάποιοι προηγουμένως. Το ψηφοδέλτιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει υποψηφίους ευρωβουλευτές, οι οποίοι θα αναλάβουν και την έδρα. Αν κάποιος είναι απλός υποψήφιος, οι ψηφοφόροι λέγουν ότι το ψηφίζουμε και αν το ψηφίζει θα πρέπει να είναι και σε θέση, θα πρέπει να είναι και πρόθυμος να ε, ασκήσει τα καθήκοντα του Ευρωβουλευτού. Σε αντίστοιχη περίπτωση να μην είναι καθόλου στο ψηφοδέλτιο. Δεν μπορούμε όμως αυτό να το δεσμεύσουμε νομικά, αλλά μπορούμε να ε, υιοθετήσουμε τη διατύπωση που προτείνει ο εισηγητής και να το υποστηρίξουμε. Τώρα για την ισορροπία του φίλου. Νομίζω είναι πάρα πολύ ασθενής η διατύπωση. Δεν θα πρέπει απλώς να διατρανώνουμε την αρχή, ε, επιτρέποντας ε, σε όλα τα κόμματα να την παραβιάζουν. Όταν μιλούμε για ισορροπία των φίλων θα πρέπει να υπάρχει ουσιαστική ισορροπία. Η Σαντρίν θα σας τα πει νομίζω αυτά περισσότερο. Κάτι άλλο. Η ενδοκομματική, η ισοκομματική δημοκρατία. Εσύ είπες ότι εμείς θα επιλέξουμε ε, τους υποψηφίους μας με προκριματικές εκλογές και είπες και καλή τύχη. Μπορεί να είναι υπερβολικά φιλόδοξο αυτό. Με ενδιαφέρει και εμένα να δω ε, ποια θα είναι η έκβαση αυτού του πειράματος. Πάντως, σε καμία περίπτωση δεν προτείνουμε αυτό να αντιγραφεί. Αν είναι αυτό πραγματικά ε, ο χρυσός κανόνας δεν είναι αυτός. Εμείς μιλούμε για μια βασική προδιαγραφή. Όλη η δημοκρατική διαδικασία, η όλη εκλογική μάλλον διαδικασία να διεξάγεται δημοκρατικά από την αρχή μέχρι το τέλος. Δημοκρατικά τι σημαίνει. Ελεύθερη, μυστική ε, ε, ψηφοφορία ε, με όρους ισότητας. Δηλαδή έχουμε ακόμα εδώ βουλευτές, συναδέλφους που εξελέγησαν πρώτα από το κόμμα τους και μετά από τους ψηφοφόρους. Αυτό θέλουμε. Και όχι ε, να είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού, παζαριού εντό του κόμματος ή γιατί έχουν έρθει εδώ λίστα επειδή ε, αρέσουν ή δεν αρέσουν στον πρόεδρο του κόμματός τους. Αυτό δεν βοηθάει ε, την νομιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ούτε προάγει τη δημοκρατία. Θα πρέπει να το λύσουμε αυτό στο ψήφισμά μας ότι ε, η όλη εκλογική διαδικασία θα πρέπει να είναι δημοκρατική, ε, με ισότητα, ελευθερία και μυστικότητα. Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο φιλόδοξοι, τουλάχιστον εμεί αυτό θα επιθυμούσαμε, αλλά γενικά να επαναλάβω ότι είναι πολύ καλή η έκθεση, μας βρίσκει σύμφωνους, όπως και όλες οι συμβαστικές τροπολογίες. Σε μερικές μόνο περιπτώσεις ζητάμε λίγο περισσότερο. Ευχαριστώ. Yes, in original... Ναι, στην αρχική διατύπωση και σε πολλές από τις ε, τροπολογίες ε, λέξεις όπως ενθαρρύνει ή προτείνει ε, χρησιμοποιούνται γιατί φυσικά τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να υποχρεωθούν ε, με κανένα τρόπο στο πώς θα προχωρήσουν και δεν μπορούμε επίσης να τους οδηγήσουμε, να τους επιβάλλουμε, να επιτρέψουν στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να έχουν τα σήματά τους ή το ονόματά τους στα ψηφοδέλτια ούτε μπορεί η Κομισιόν να επιβάλλει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία επισήμω. Αυτό που θα ήθελα να γνωρίζω και αυτό δεν το καταλαβαίνω ούτε από την αρχική διατύπωση ούτε και από τις τροπολογίες είναι αν προβλέπετε πως αυτά τα ευρωπαϊκά πολιτικά ή μάλλον οι εκπομπέ των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων θα είναι αντί για την τροπολογία και η τροπολογία 56 το υπονοεί αυτό αν θα είναι σε αντικατάσταση και όχι σε συμπλήρωση ή παράλληλα με τις εκπομπές των εθνικών ε, πολιτικών κομμάτων. Έπειτα τα ονόματα και τα ε, σήματα θα είναι επίσης σε αντικατάσταση των εθνικών πολιτικών κομμάτων ή θα εμφανίζονται και τα δυο ε, σήματα ή εμβλήματα των δυο εθνικού και ευρωπαϊκού κόμματος. Και έπειτα η Κομισιόν φαίνεται να έχει φτιάξει ένα ευφιέστατο ε, πρόγραμμα γιατί ακολουθεί τα όσα γίνονται στις ε, κοινοβουλευτικές δημοκρατίες από τη στιγμή που αναπτύχθηκαν ε, τα πολιτικά κόμματα τον 19ο αιώνα οι κοινοβουλευτικές εκλογές σιγά σιγά μετατράπηκαν σε πρωθυπουργικές εκλογές όπως είναι σήμερα και είναι πολύ ευφιές όπως είπα αυτό το σχέδιο όμως είμαι πεπισμένος πως στο εγγύς μέλλον οι ψηφοφόροι θα γνωρίζουν ελάχιστα για την Κομισιόν και τις λειτουργίες τους και ακόμα λιγότερα για τους διάφορους υποψηφίους ιδιαίτερα αυτούς που προέρχονται από άλλα κόμματα εκτός του δικού τους. Δεν θέλω να φανώ κακός, ε, αλλά εγώ προσβλέπω σε ένα βαθμό σύγχυσης και χάους. Φυσικά αν λειτουργήσει και αν υποψήφοι ας του κόμματος Α κερδίσουν ε, τις ψήφους που χρειάζονται, θα ιτηθούν από όλα τα άλλα κόμματα. Ο κύριος Μορέιρα, νομίζω στην τροπολογία 70, λέει, προτείνει μάλλον το κόμμα που θα έχει πολλές ε, έδρες και ψήφους θα πρέπει να είναι η πρώτη επιλογή. Αλλά ακόμα και αυτή η τροπολογία δεν προχωρά μέχρι του να πει ότι θα είναι η ίστατη λύση, η ίστατη επιλογή, άρα θα είναι πιθανόν ε, το κόμμα που θα έχει κερδίσει τις περισσότερες έδρες και ψήφους να μην έχει τον υποψήφιό του ως ε, επίτροπο. Τώρα όσον αφορά τις ισορροπίες φύλου, όλα αυτά ακούγονται πολύ υπέροχα και, με, θα, και εγώ θα ήμουν πολύ ικανοποιημένος αν κάθε κοινοβούλιο στον κόσμο έχει περίπου μια ισορροπία ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες βουλευτές ή ευρωβουλευτές για το Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά αν τα κόμματα είτε θελοντικά είτε υποχρεωτικά έχουν ίσους αριθμούς με τη βάση του κριτηρίου του φύλου, αυτό δεν είναι κάτι πλέον που δεν κοστίζει τίποτα. Αυτό γίνεται εις βάρος άλλων κριτηρίων, που σημαίνει ότι τα δύο κριτήρια της αξίας, της ικανότητας δηλαδή να κάνει κανείς τη δουλειά του και το άλλο κριτήριο της πολιτικής άποψης μέσα στο πλαίσιο του συγκεκριμένου πολιτικού κόμματος θα έρθουν ε, δεύτερα. Και αυτό νομίζω πως είναι πολύ ψηλό ως τίμημα. Ευχαριστώ πολύ. Το δικό μου σχόλιο είναι πως η πολιτική, ε, μάλλον η αξία και η πολιτική γνώμη ισχύουν το ίδιο και για άνδρες και για γυναίκες, οπότε δεν βλέπω κανένα πρόβλημα. Η Σαντρίν Μπελιέ τώρα. Να ακούσουμε. Ευχαριστώ στα σχόλιά σα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επιτρέψατε μου να κάνω μια παρατήρηση καταρχήν. Βρίσκω πως είναι κρίμα και ότι είναι και λυπηρό ε, και δύσκολα καταλαβαίνω το κοινοβούλιο μας και η Επιτροπή μας προβλέπει να συζητήσει τις αρμοδιότητες της για να καθορίσει ε, και να ορίσει την έδρα του ή και το χρονοδιάγραμμα εργασίας του, ενώ ταυτόχρονα αρνείται την πρόταση διοργάνωσης των εκλογών που στόχο έχουν να ενισχύσουν τη συμμετοχή και τον εκδημοκρατισμό του Κοινοβουλίου μας αλλά και την εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λυπούμε λοιπόν ε, σε αυτό το στάδιο για την ελαφρότητα και τις απόφασεις που ελήφθη στη διάσκεψη των Προέδρων. Ήθελα να ξεκινήσω με αυτή την παρατήρηση. Επίσης ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όπως και οι άλλοι ομιλητές τον Άντριου Ντάφ, τον εισηγητή για την εργασία του. Να τον ευχαριστήσω επίσης ε, διότι δεν απέρριψε τις, τροπολογίε τις ε, τροπολογίες που υπέβαλα καθυστερημένα και ευχαριστώ εκ των προτέρων τα μέλη της Επιτροπής που ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση και έπειτα όπως και το θύμισε και εκείνος ε, αυτή η έκθεση τίνει να εθαρρύνει τα ευρωπαϊκά κόμματα να υποβάλουν υποψήφιους για την Προεδρία του Κομισιόν. Ήταν μια από τις καινοτομίες, ένα από τα στοιχεία που μπορεί να επιτρέψουν να ξανα να, να εκδημοκρατιστεί, να δοθεί εμπιστοσύνη, να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη και να δημιουργηθεί νόημα και ενδιαφέρον για τους Ευρωπαίους εκλογείς τη στιγμή που θα εκλέξουν τους ε, βουλευτές τους. Για να βελτιωθεί η ποιότητα λοιπόν της εκστρατείας των ευρωεκλογών, να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή και να ενθαρρυνθεί βεβαίως και η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκστρατεία που θα γίνει σε κάθε κράτος. Εμείς θα στηρίξουμε τις, εισηγη... τις συμβαστικές που έφτιαξε ο εισηγητής. Είναι καλή ισορροπία ενώ παραμένει φιλόδοξο το προσχέδιο. Ήθελα απλώς να επιμείνω και πάλι στις προτάσεις που εγώ επέβαλα ώστε να εξασφαλιστούν οι στόχοι που αναφέρθηκαν ε, για τέσσερα τουλάχιστον σημεία. Καταρχήν για το στόχο της ισότητας των ε, ψηφοδελτίων σε εθνικό επίπεδο πιστεύω πως θα έχουμε λιγότερες δυσκολίες ή εν πάση περιπτώσει πως θα είναι λιγότερο δύσκολο να εξασφαλίσουμε την ισότητα από ότι να εξασφαλίσουμε το στόχο οι υποψήφοι στο Ευρωκοινοβούλιο να ε, να ολοκληρώσουν τη θητεία τους στο Ευρωκοινοβούλιο από τη στιγμή που θα έχουν εκλεγεί. Πιστεύω λοιπόν ότι κάθε κράτος και κάθε κόμμα θα έχει λιγότερη δυσκολία να βρει ε, ε, να τηρήσει μάλλον την ισότητα, να βρει υποψηφίους άντρες και γυναίκες, παρά να βρει ανθρώπους που θα τηρήσουν, θα ολοκληρώσουν τη θητεία τους. Για την υποψηφιότητα στην ε, Κομισιόν πιστεύω πως είναι ενδιαφέρον να συνεχίσουμε να καλούμε το σύνολο των ευρωπαϊκών πολιτικών ε, κομμάτων να κάνουν ε, ε, εκλογές. Μάλιστα οι πράσινη αυτό αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε. Θα το κάνουμε αυτό και έχουμε κάθε ελπίδα να το υλοποιήσουμε. Για το άνοιγμα των εθνικών ψηφοδελτίων σε Ευρωπαίους υποψηφίους ε, δεν, δεν το έχουμε κάνει αυτό δεν, ε, ε, ε, δεν είναι η πρώτη φορά. Το 2009 είχαμε πρώτον τον Ντανιέλ Κονμπεντίτ που είναι γερμανικής υπηκοότητας και στηρίζουμε οτιδήποτε μπορεί να γίνει για να κατευθυνθούμε προς αυτήν την πορεία ώστε να δοθεί περισσότερη ευρωπαϊκή διάσταση σε αυτές τις ευρωεκλογέ. Και έπειτα ανάμεσα στι τροπολογίες μου επανήλθα σε αυτή την ανάγκη διοργάνωση συζητήσεων ανάμεσα στους υποψηφίους των διαφόρων πολιτικών κομμάτων, ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων που έχουν υποψήφιους για το πρόεδρο της Κομισιόν. Ξέρουμε ποιος είναι ο ρόλος της τηλεόρασης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης και αν μπορούσαμε τουλάχιστον δύο-τρεις συζητήσεις να διοργανώσουμε σε όλες τις γλώσσες και να ε, παρουσιαστούν από όλες τις, τις δημόσιες τηλεοράσεις ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη κινητοποίηση για αυτές τις εκλογές. Και έπειτα κάτι ακόμα το οποίο στηρίχθηκε και από άλλες πολιτικές ομάδες είναι το γεγονός ότι επιβεβαιώνουμε ακόμη μια φορά την σημασία στην επόμενη αυτή εκλογική εκστρατεία των, ευρω... των πραγματικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, των βάσεων, αυτό που λέει ο Ρούντολφ, πλατφόρμες και ότι το σύνολο των εθνικών πολιτικών κομμάτων να ιδιοποιηθούν και να αναλάβουν αυτά τα προγράμματα για αυτές τις ευρωεκλογέ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Άντριου Ντάφ σαφώς είπε ότι θα ήθελε να έχει την έγκριση της Επιτροπής για τις τροπολογίες που έφτασαν καθυστερημένα. Ε, να, να σας ρωτήσω, συμφωνείτε? Εάν δεν υπάρχει αντίρρηση, βεβαίως ε, γίνονται δεκτές οι τροπολογίες σας. Ε, αφού κάναμε και την ε, διαδικασία που έπρεπε. Ο Άντριου. Ευχαριστώ πολύ όλους όσους πήραν το λόγο και όλους όσους θα μπορούσαν να, ε, να μην μιλήσουν, να μιλήσουν αλλά δεν μίλησαν, γιατί και αυτό βοηθάει πολύ συχνά. Κατανοώ την ανησυχία του ΕΛΚΑ και των Σοσιαλιστών σε σχέση με την τροπολογία 69 και όλα αυτά. Και θα κάνω μια προφορική τροπολογία που θα διευκρινίσει τα πράγματα και που θα μας βάλει στο σωστό δρόμο αλλά πάντως είναι σωστό ως αύκο να, εμείς να παροτρύνουμε, να προωθούμε την διάσκεψη των Προέδρων ώστε να ξεκινήσει να κάνει πια δουλειά, να βρει μια συμφωνία όπως ε, μας ε, ζητά να κάνουμε και η συνθήκη ανάμεσα σε εμά και το Συμβούλιο για τις λεπτομέρειες της ε, συμβουλευτικής διαδικασίας που θα ακολουθήσει τις εκλογές. Και ε. αυτό θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί και να έχει γραφτεί το τι θα γίνει. Εγώ δεν εμπιστεύομαι μια προφορική συμφωνία ανάμεσα στον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου και τον πρόεδρο του Συμβουλίου. Για το τι θα συμβεί μετά. Από εμά εξαρτάται νομίζω να επιμείνουμε. κοινή συνενέση όπως ορίζει και η συνθήκη. Αυτό θα το αναφέρω σε μια τροπολογία αύριο. Και θα κοιτάξω ξανά και την συμβαστική έξι ώστε να είμαι βέβαιος, ε, 7 με συγχωρείτε, για να είμαστε σίγουροι για το τι ακριβώς λέει. Τώρα, για τον ε, Ράφαλ Ταρσκόφσκι που μιλά για που μίλησε για αυτή την ιδέα του να αναμένουμε ότι ο υποψήφιος θα αναλάβει τη θέση του Ευρωβουλευτή από τη στιγμή που έχει μπει υποψήφιος. Θυμάμαι ότι το προηγούμενο Νοέμβριο περάσαμε ένα ψήφισμα που ζητούσε τουλάχιστον το 50% του συνόλου των επιτρόπων να προέρχεται από ευρωβουλευτές. Είναι πολύ ψηλό το ποσοστό και θα με εντυπωσίαζε αν το καταφέρναμε. Αλλά το προηγούμενο της εκλογής ενός ευρωβουλευτή που εκλέγεται την Άνοιξη και έπειτα μεταγράφεται το φθινόπερο στην Κομισιόν είναι κοινό. Ο Μισελ Μπαρνιέ είναι ένα παράδειγμα. Ο Λεβαντόφσκι και εκείνο νομίζω. Και αυτό αυξάνει την νομιμότητα του ίδιου του Επιτρόπου. Αφού έχουν προηγούμενα εκλεγεί σαν ευρωβουλευτές. Θα πρέπει να επιμείνουμε λοιπόν σε αυτό που θέλουμε εδώ και να βρούμε μια διατύπωση που να λειτουργεί. Και συμφωνώ απόλυτα με τον Τζέρελτ ότι το βασικό είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι υποψήφοι για την Προεδρία της Κομισιόν θα είναι δημοκρατικά θεμητοί σε αυτό συμφωνούμε. Ο τρόπος είναι πόσο, πόσο δηλαδή περιγραφική θα μπορούμε να είμαστε σε αυτή τη φάση, σε αυτό το ψήφισμα. Στον κύριο Μπρόντζ, Εγώ θεωρώ πως ε, οι εκπομπές των εθνικών ε, πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών ε, πολιτικών κομμάτων στη τηλεόραση θα είναι παραπληρωματικές. Δεν θα είναι η μία προς αντικατάσταση της άλλης. Το ίδιο και για τα ονόματα ή τα εμβλήματα. Θα πρέπει να, πρέπει να δούμε και τα δύο. Όσο γίνεται πιο κοντά το ένα στο άλλο, στις αφήσει αλλά και στα ψηφοδέλτια. Και όπως είπε και ο κύριος Μπρόντς, για το πώς ακριβώς γίνεσαι πρόεδρος της Κομισιόν, σίγουρα βέβαια χρειάζεται να σε προτείνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και ο κύριος Μορέιρα πρότεινε καταρχήν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εξετάζει το, να βλέπει μάλλον ποιο πολιτικό κόμμα έχει τις περισσότερες έδρες στο Κοινοβούλιο. Αλλά στη συνέχεια η συνθήκη είναι απόλυτα σαφής ότι το εν λόγω άτομο θα μπορεί να αναλάβει αυτή τη θέση του Προέδρου της Κομισιόν αν έχει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου. Αν αυτό δεν συμβεί δηλαδή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να αναζητήσει έναν δεύτερο υποψήφιο, που ίσως να μην είναι από το μεγαλύτερο κόμμα, αλλά από κάποιο συνασπισμό, από κάποια συνένεση διακομματική που ίσως στο τέλος να μπορεί να επιτύχει και να είναι και πρόεδρος μεγαλύτερου βεληνικούς. Δεν ξέρω, είναι ένα πείραμα. Και για να είμαστε σαφείς για το πόσο πειραματικοί η ε, ε, φαντεζοί θα είμαστε σε αυτή την εκλογική εκστρατεία, συμφωνώ απόλυτα με τη Σαντρίν Μπελιέ ότι ότι θα πρέπει να υπάρχει ισότητα ανάμεσα ότι θα πρέπει να γίνουν συζητήσεις ανάμεσα στους υποψηφίους και το έχω συμπεριλάβει και αυτό στην πρότασή μου. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ε, I strongly... ευχαριστώ. Είναι όντως κρίσιμο διότι υπήρξε μεγάλη αποχή στις Προηγούμενε ευρωεκλογέ. Θα χρειαστούμε λοιπόν καλούς υποψηφίου και συζητήσει και ίσω έχουμε την ευκαιρία έτσι να φέρουμε κοντύτερα την Ευρώπη στις και στου πολίτες μας, διότι ω γνωρίζετε υπάρχει μεγάλο έλλειμμα. Και μέσα βέβαια σε αυτή την οικονομική και κοινωνική κρίση, θα έλεγα και δημοκρατική. Καλώς ήρθατε αγαπητοί κύριοι για την ακρόαση γνωρίζετε ότι θα διεξαχθεί ψηφοφορία αύριο και είμαι βεβαία ότι θα είστε όλες και όλοι εδώ για να έχουμε την απαραίτητη απαρτία. Ακολουθεί ο προϋπολογισμός 2014. Πρέπει να μιλήσουμε και για την εντολή για τριμερή διάλογο. Ο κύριος Μέσσερ Σμιτ έχει τοποθετηθεί σχετικά αντιπρόεδρος για την προηγούμενη, στην προηγούμενη μάλλον συνεδρίαση. Έχουμε λάβει ως γραμματεία δηλαδή 22 τροπολογίες από ορισμένους βουλευτές uh, uh, και από τον ίδιο τον εισηγητή. Μας μένουν τώρα πριν από την ακρόαση 15 λεπτά. Παρακαλώ λοιπόν τον εισηγητή να κάνει την εισαγωγή στην γνωμοδότησή του και, την, και τις προτινόμενες συμβαστικές τροπολογίες. Ελπίζω και ορισμένες ή ορισμένοι συνάδελφοι να κάνουν σχόλια. Παρακαλώ να σηκώνετε καλά τα χέρια. Ελπίζω να έχουμε... Έχετε λοιπόν το λόγο κύριε Σιγητά. Ναι, θα είμαι σύντομος. Έχουμε ήδη εξαγάγει σχετική συζήτηση και όλοι έχουν κάνει τις τροπολογίες τους. Είναι δύσκολο να επιτευχθεί συμβασμός επί των τροπολογιών αυτών, από τις οποίες ορισμένες δεν περιορίζονται μόνο στο θέμα της γνωμοδοτήσεως, αλλά ξεφεύγουν προς πάσα κατεύθυνση. Εγώ προτείνω λοιπόν απλώς να τις ψηφίσουμε αύριο. Όλες και όλες 22 είναι. Δεν είναι δύσκολη η ψηφοφορία αυτή. Έχω ήδη διανύμει τις προτιμήσεις μου για το πώς να ψηφίσουν διάφορες, να ψηφιστούν μάλλον διάφορες τροπολογίες. Εγώ δεν έχω άλλο τίποτε να προτείνω. Έχω ήδη διανύμει την πρότασή μου, όπως σας είπα. Έχω αποστείλει και πρόσκληση για συνάντηση μεταξύ εμού και των σκιωδών εισηγητών, οι οποίοι δεν ανταπεκρίθηκαν, ανταπεκρίθησαν ναι, ελπίζω οι συνάδελφοι να προσπαθήσουν να βελτιώσουν το κείμενο. Χέφνερ, ναι, ευχαριστώ. Ένα θέμα θέτω, αλλά καλύτερα στα γερμανικά. Γενικά νομίζω οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σμιτ για την γνωμοδότηση του. Εμάς μας ικανοποιεί και θα την υπερψηφίσουμε. πολιτικέ διαφορέ περιορίζονται στην τελευταία παράγραφο. Υπάρχουν όμω και πολλέ τροπολογίε σχετικά για τι οποίε θα ψηφίσουμε αύριο. Άρα δεν θα υπησέλθω σήμερα σε λεπτομέρειες τη συζήτηση. Πρόκειται για θέμα πολιτική αξιολογήσεω. Η δική μα πολιτική αξιολόγηση είναι διαφορετική από αυτήν του εισηγητού. Θεωρώ ότι και η πλειοψηφία της Επιτροπής θα δει το θέμα όπως εμείς. Ένα θέμα θέλω να τονίσω. DCI. Και μιλώ για την ε, πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών που εισήχθη χωρίς να υπάρχει το απαραίτητο πλαίσιο. Η ιστοσελίδα της Κομισιόν δεν λειτουργούσε πριν ένα πεντάμινο, κάτι το οποίο οδήγησε σε μεγάλη απογοήτευση πολλών και δυσαρέσκεια. Τώρα λειτουργεί ως τούτο λύση μέσω ενός hosting στο Λουξεμβούργο προσωρινά. Κοιτάξτε, η διαδικασία αυτή, αυτή η μεγάλη προσφορά προς τους Ευρωπαίους πολίτες αμφιωτέρων των φίλων να μπορούν να εκφράσουν δηλαδή άποψη, να κάνουν προτάσεις ε, στους φορείς της Ένωσης. Δεν μπορεί λοιπόν να αντιμετωπιστεί με τέτοιες πρόχειρες εμβαλωματικές λύσεις οι οποίες δεν είναι και γερά θεμελιωμένες στο δίκαιο. Δεν έχουν τον απαραίτητο προπολογισμό ούτε το απαραίτητο στελεχικό δυναμικό. Άρα πρέπει να οργανωθεί καλύτερα η Κομισιόν. Γι' αυτό και θεωρούμε απαραίτητο να οργανωθεί καλύτερα η ανταπόκριση αυτή, όπως ζητεί και ο εισηγητής, και ο προπολογισμό να αυξηθεί και η πρωτοβουλία να είναι σε θέση να διατυπωθεί καλύτερα, αλλά ιδίω στην Κομισιόν να υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα, δηλαδή κονδύλια, προσωπικό, ώστε να μπορούν να διατυπώσουν καλά και γρήγορα την διαδικασία, να προχωρήσουν τη διαδικασία, να δώσουν συμβουλές στους πολίτες, να κάνουν την διοικητική επεξεργασία της ε, πρωτοβουλίας και το Europe Direct να εκπαιδευτεί καθώς και άλλες υπηρεσίες της Κομισιόν, ώστε στο μέλλον να μπορούν να ανταποκρίνονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Υπάρχει, όπως είπα, μεγάλη δυσαρέσκεια και απογοήτευση από πλευρά των πολιτών και γι' αυτό είναι απαραίτητο να γίνουν τα βήματα αυτά. Παρακαλώ λοιπόν να υποστηρίξετε την τροπολογία μας. Κατά τα άλλα, εμείς υποστηρίζουμε τις προτάσεις που έχουν γίνει. Ευχαριστώ κύριε ε, συνάδελφε. Εσείς τώρα κύριε Αντιπρόεδρε Φόξ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο κύριο Μέσσερ Σμιτ για την γνωμοδότησή του. Και μου αρέσει πολύ που λέει να μειωθεί το γραφειοκρατικό κόστος εντός της ενώσεως. Δεν τα βλέπει κανείς συχνά αυτά και είμαι βέβαιος ότι οι συνάδελφοί μου θα καταψηφίσουν τη σχετική του πρόταση γιατί εδώ συνήθως προτιμούν να αυξάνονται οι προπολογισμοί και όχι να μειώνονται. Επίση μου αρέσει το γεγονό ότι ο φίλο Μέσο Σμιτ σχολιάζει επί του προβλήματο που αντιμετωπίζουμε με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Αν είχα επιλογή, εγώ δεν θα άφηνα χρηματοδοτηθεί κανένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, διότι είναι πεταμένα λεφτά των φορολογουμένων. Κάποια λεφτά βεβαίω θα δαπανηθούν σε πολιτικά κόμματα. Είναι λάθο, λοιπόν να μπούμε στο παιχνίδι αυτό όπου το Κοινοβούλιο αποφασίζει ποια κόμματα είναι αποδεκτά και ποια όχι. Κάτι τέτοιο είναι πολύ επικίνδυνο και πολύ φοβούμαι ότι θα οδηγήσει σε ε, πολύ κακή φήμη του Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ τον κύριο Μεσέσουμιτ για την έκθεσή του. Ευχαριστώ κύριε Μπρόνξ και να ολοκληρώσουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και σε άλλα θέματα. Ναι, παράγραφος 5 της εκθέσεως καταδικάζει ως αντιδημοκρατικό δημοκρατικό, δημοκρατική πάσα προσπάθεια να γίνει επιλογή μεταξύ των κομμάτων. Αυτά τα έχει πει βέβαια ο κύριος Μέσο Σμιτ και ο κύριος Φόξ. Ο κύριος Νταφ απάντησε για το εάν τα πολιτικά μηνύματα των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων θα είναι συμπληρωματικά ή υποκατάστατα, ότι θα είναι συμπληρωματικά. Δεν πρόκειται λοιπόν τόσο πολύ για διάκριση μεταξύ ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, αλλά διάκριση κατά εθνικών πολιτικών κομμάτων σε ευρωεκλογέ. Διότι αναλογικά θα λαμβάνουν λιγότερο χρόνο, αν κατάλαβα καλά από αυτά που είπε ο κ. Νταφ. Ναι. Αυτό είπε. Πράγματι, ορίστε, συμφωνεί. Ναι. Θα ρωτήσω τον εισηγητή αν επιθυμεί να κάνει κάποιο σχόλιο ακόμη. Ναι, σας ευχαριστώ κύριε Σιγήρη για τα σχόλια. όντως υπάρχει κάποια διαφωνία επί θεμάτων μεταξύ του CRE από εδώ και των υπολείπων από την άλλη. Εγώ προσπάθησα να τάμω με ρεαλιστικό τρόπο και γι' αυτό τροποποίησα και δική μου πρόταση. Αλλά στο πνεύμα της συνεργασίας, έτσι, κινήθηκα εγώ και ελπίζω οι συναδελφοί μου να το εκτιμήσουν. Αυτά για την παραγραφό 5 για το 4, κύριε Χέφνερ, η δική μου πρόταση είναι να υποστηριχθεί η τροπολογία του κύριου Χέφνερ. Δεν βλέπω λοιπόν κανένα πρόβλημα εδώ. Και στον τομέα ειδικά αυτό, θεωρώ ότι είναι τεχνικό πρόβλημα το, αυτό το οποίο τονίζω στην παράγραφο 4 και νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει γενικότερη προσέγγιση, αυτή δηλαδή της παράγραφου 7. Δεν βλέπω πού να διαφωνήσουμε. Ακριβώς για αυτό το λόγο δε παρετήθηκα από κάθε ιδέα συμβασμού. Βρίσκω ότι είναι και απλούστερο και δημοκρατικότερο να ψηφίσουμε. Ευχαριστώ λοιπόν για τις διάφορες ιδέες που καταθέσατε και αναμένω την πορεία της ψηφοφορίας αύριο. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Όπως είπα πριν, αλλά επειδή ήταν ορισμένοι απόντες πριν, για την κατανομή των εδρών όπως ζητήθηκε και για σας κύριε Φόξ πρόκειται γι' αυτό θα ψηφίσουμε αύριο στις 10 και 35 όπως συμφωνήθηκε στην αρχή της συνεδριάσεώς μας και όλα τα υπόλοιπα μετά ευχαριστώ λοιπόν τώρα σας παρακαλώ τρία λεπτά διάλειμμα και αμέσως μετά θα αρχίσουμε την ακρόασή μας που τη βρίσκω εξαιρετικά σημαντική. Θα συνεχίσουμε λοιπόν σε τρία λεπτά. Okay, so dear colleagues, the three minutes is over. Πέρασαν τα τρία λεπτά. Έχω το, έχω το θλιβερό καθήκον να σας ε, υπομνήσω ότι τελείωσαν τα τρία λεπτά το διάλειμμα δηλαδή, αγαπητές κυρίες και κύριοι, και επομένως... Αλλά τώρα δεν έχει μικρόφωνο πλέον η κυρία Γκουρμάη. Okay. Καλά λοιπόν. Σας ευχαριστώ για την υπόμονή σας. Και βεβαίως με τον τρόπο αυτό δείχνουμε και στους εμπειρογνώμονες μας ότι τηρούμε με ακρίβεια το χρονοδιάγραμμα. Όπως είπα, πιστεύω ότι η ακρόαση είναι σημαντική. Έχει σχέση με το δικαίωμα αυτοδιοργάνωσης των εργασιών του Κοινοβουλίου με στόχο να ενισχύσουμε τον προβληματισμό γύρω από το δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να οργανώσει τον τρόπο εργασίας του όπως προκύπτει από το 232 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε λοιπόν τους εξής εμπειρογνώμονες. Θα πω λίγα για το βιογραφικό του καθενός που νομίζω ότι είναι σημαντικό για να ξέρουμε όλοι ποιον έχουμε μπροστά μας. Έχουμε πρώτα τον κύριο Ολιβιέ Κώστα, καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Μπορντό και ανώτερο στέλεχος ερευνητή του Εθνικού Κέντρου Ερευνών και επισκέπτη καθηγητή στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελών, στο Κολέγιο της Ευρώπης και στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης. Ο κύριος Κώστα έχει συντάξει πολλά στάνταρ έργα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ιδιαίτερα και είναι υπεύθυνο για το τμήμα Ευρωπαϊκών Σπουδών του Γαλλικού Συνδέσμου Πολιτικών Επιστημόνων και μέλος του Συντακτικού Συμβουλίου του περιοδικού της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Με πολλές δημοσιεύσεις, δημοσιεύσεις δεν θα σας διαβάσω όλες, άλλωστε είναι δημοσιευμένες οι δημοσιεύσεις και μπορείτε να διαβάσετε και πολλές βέβαια σχετικά με το Κοινοβούλιο, την συναπόφαση και τον εγχώριο νομοθέτη, καθώς βέβαια και την ανανέωση του κοινοβουλευτισμού στην Ευρώπη και λοιπά Αυτά θα τα δείτε, όπως είπα. Άρα, θαυμάσιο πλαίσιο όπου εργάζεστε κύριε, σας παρακαλώ να προβείτε στην διάλεξή σας. Έχετε δέκα λεπτά, όπως θα γνωρίζετε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως γνωρίζω είναι πολύ πιο εύκολο για τους διερμηνείς να, να μιλήσει κανείς στη μητρική του γλώσσα, γι' αυτό και θα μιλήσω γαλλικά. Je vais me prononcer surtout sur la question de, de l'autonomie organisationnelle du Parlement. Θα μιλήσω για την αυτονομία, την οργανωτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κοινοβουλίων εν γέννη. Θα πρέπει νομίζω να προχωρήσουμε σταδιακά για να κατανοήσουμε καλά τα πράγματα. Καταρχήν, θα πρέπει να πούμε δύο λόγια για το τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ω πολιτικό σύστημα. Και για να ε, φέρουμε άποψη, θα πρέπει να μιλήσουμε για μια πρώτη δυσκολία, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ω πολιτικό σύστημα είναι το αποτέλεσμα ενό. Ε, συμβιβασμών ε, μιας ε, δαρβενικής διαδικασίας που δεν είχε κάποιο προκαθορισμένο σχήμα, δεν βασίστηκε σε κάποια συγκεκριμένη πολιτική θεωρία και δεν έχει ε, ούτε και αποστεριώρη πολιτική θεωρία, γιατί είδαμε ότι η σύμβαση για την Ένωση, η συνέλευση για την Ένωση δεν μπόρεσε να καταλήξει σε συγκεκριμένε ε, απλές αξίες για να εξηγήσει το ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα, το σύστημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενισχύθηκε το Ευρωκοινοβούλιο Διαρκώ. η συνθήκη λέει άλλα πράγματα από ό,τι έλεγε στην δεκαετία του 50 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λέει επίση πω η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή τη δημοκρατική εκπροσώπησης, αλλά όταν το λέει αυτό το Ευρωκοινοβούλιο Κοινοβούλιο αλλά και την έμεση εκπροσώπηση των πολιτών στο, Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τελειώνει μάλιστα αναφέροντα ε, την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Όλα αυτά είναι αρκετά συγκεχημένα. Υπάρχει δηλαδή ένα πολιτικό σύστημα κάπω μυστήριο, δύσκολο να θεωρητικοποιηθεί και είναι και δύσκολο να κατανοήσει κανεί το καθεστώ του Ευρωκοινοβουλίου και μέσα σε όλη αυτή την υπόθεση. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι το Ευρωκοινοβούλιο εξακολουθεί να μην, καθο... να μην ορίζεται ω κυρίαρχη ε, συνέλευση. Δεν έχουμε άρθρο όπω έχουμε στα διάφορα συντάγματα το Κοινοβούλιο που να λέει ότι το Κοινοβούλιο εκπροσωπεί το λαό και άρα πρέπει να αποφασίζει για όλα τα πράγματα. Η συνδίκη λέει πω το Κοινοβούλιο πρέπει εν γέννη να συνδέεται στι νομοθετικέ και δημοσιονομικέ διαδικασίε και στον έλεγχο, αλλά μέχρι εκεί. Ε, επίση, οι σχέσει του Ευρωκοινοβουλίου με τα άλλα θεσμικά όργανα είναι κάπω παράξενε ε, ανάμεσα σε ένα προεδρικό σύστημα και ένα κοινοβουλευτικό σύστημα. Όλα αυτά δεν είναι πολύ σαφή. Οι συνθήκε δεν είναι επίση σαφεί όσον αφορά βαθμό αυτονομία του Ευρωκοινοβουλίου. Έχουμε ένα μεγάλο βαθμό αυτονομία του Ευρωκοινοβουλίου που βασικά όμω είναι ιστορικό ατύχημα. Ε, επειδή στην αρχή το Ευρωκοινοβούλιο δεν είχε καμιά εξουσία, οι συντάκτες των συνθηκών δεν χρειάστηκε να υποχρεώσουν αυτό εδώ το, σύστημα, το θεσμό ώστε να το περιορίσουν, ε, να περιορίσουν την οργανωτική του αυτονομία ή να το αναγκάσουν να λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο. Και γι' αυτό και απορρέει, από αυτό απορρέει η αυτονομία του Ευρωκοινοβουλίου όσον αφορά την εσωτερική του διοργάνωση, τον αριθμό των επιτροπών, την ατζέντα και για όλα αυτά το Ευρωκοινοβούλιο έχει πολλές ελευθερίες. Αυτό που είναι επίση αξιοσημείωτο είναι ότι το Συμβούλιο και η Κομισιόν ποτέ δεν αμφισβήτησαν αυτή την αυτονομία. Πολύ λίγε προσφυγέ έγιναν κατά των αποπειρών του Κοινοβουλίου να επεκτείνει τι εξουσίε του ε, και να ξεπεράσει ακόμα και το γράμμα των συνθηκών. Ενώ θα μπορούσε κανεί να φανταστεί πως κανονικά το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα αφισβητούσαν αυτέ τι θεσμικέ στρατηγικέ του Κοινοβουλίου. Και επίση ε, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεν μπορούν να ασκήσουν πολιτική πίεση δεδομένου των πολιτικών κομμάτων και πώς αυτά λειτουργούν μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Το μόνο πραγματικό όριο στην αυτονομία του Ευρωκοινοβουλίου είναι βεβαίω η έδρα και το χρονοδιάγραμμα που συνδέεται με το θέμα της έδρας διότι η συνθήκη λέει πως το Κοινοβούλιο οφείλει να διοργανώνει 12 εβδομαδιαίες ολομέλειες, συνόδους ολομέλειες στην έδρα του που είναι το Στρασβούργο. Να θυμίσω ωστόσο πως η συμβιβαστική, το συμβιβασμό του Εδιμβούργου δεν επευλήθη από τις κυβερνήσεις, αλλά συμπεριλαμβάνει και την ψηφοφορία του Ευρωκοινοβουλίου για την έκθεση Πίτερς, όπως ονομάζεται, για τον Απρίλιο του 1991. Το Ευρωκοινοβούλιο εκφράστηκε στην ολομέλειά του για το θέμα της έδρας, απαντώντας σε εντάσεις που ήδη είχαν προκληθεί μέσω μιας έκθεσης για την σκοπιμότητα κατασκευής κτίριων στην, στις Βρυξέλλες. Πώς μπορούμε λοιπόν να ερμηνεύσουμε αυτή την αυτονομία του Ευρωκοινοβουλίου. Μπορούμε να έχουμε δύο εικόνες, δύο απόψεις που είναι ριζικά αντίθετες. Η μία είναι να θεωρήσουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας διεθνής οργανισμός, όχι και πολύ διαφορετικός από τους άλλους, οπότε λέμε ε, τότε πως τα κράτη-μέλη πρέπει να ορίσουν πώς θα λειτουργεί αυτός ο οργανισμός ε, συμπεριλαμβανομένες της έδρας των θεσμών του. Είναι περίπου το, άρθρο, το άρθρο 341 που λέει ότι τα κράτη-μέλη αποφασίζουν ποιο εδρεύει πού. Έπειτα μπορεί από την άλλη πλευρά να δούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως, εν, ως ένα ομοσπονδιακό κράτος και εκεί απορρέουν δυο. Από αυτό δύο προσεγγίσεις. Είτε μιλάμε για την αρχική ε, ε, ε, περιχαράκωση και να έχουμε ένα είδος κεκτημένων εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην αρχή αυτό δεν πιάστηκε, δεν περιχαρακώθηκε καθόλου και οι συντάκτες των συνθηκών άφησαν τους βουλευτές να ρυθμίσουν οι ίδιοι, να αποφασίσουν για το πού θα εδρεύουν, πώς θα λειτουργεί το σώμα, πόσες θα είναι οι εσωτερικές επιτροπές και οι εσωτερικές διαδικασίες, ο εσωτερικός κανονισμό. Και μπορεί να υπερασπιστεί το ότι αυτή ιστορική κατάσταση δημιούργησε το δικαίωμα για το Κοινοβούλιο να έχει αυτή την αυτονομία και αυτή η αυτονομία είναι και ιδρυτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και οδηγεί όντως το Ευρωκοινοβούλιο να είναι πολύ ανεξάρτητο όσον αφορά την οργάνωσή του, τον προϋπολογισμό του, τη διοίκησή του το διοικητικό του μηχανισμό. Και άρα και το θέμα της έδρας εδώ είναι κάπως ε, μια εξαίρεση που δύσκολα μπορεί κανείς να αιτιολογήσει. Ένας άλλος τρόπος να δει, αρχικά, να δει κανείς το θέμα είναι ότι η αρχική αυτή η ε, έλλειψη ότι δηλαδή τα κράτη-μέλη αρχικά δεν θεώρησαν απαραίτητο να πλαισιώσουν την τάδε δίνα λειτουργία του Ευρωκοινοβουλίου ενώ παραμένουν ελεύθερα να παρέμβουν στην λειτουργία του Ευρωκοινοβουλίου ιδιαίτερα για το θέμα της έδρας όπως το έπραξαν στον συμβιβασμό του Εδιμβούργου. Και από αυτή την άποψη θα λέγαμε ότι σε πολύ λίγα πολιτικά καθεστώτα μπορούμε να, να, να βρούμε ένα κοινοβούλιο το οποίο μπορεί μόνο να αποφασίζει για την έδρα του και εν γέννη. Η, ο ε, χώρος συνόδου του κοινοβουλίου ορίζεται από το, από το Σύνταγμα, είτε από κάποιο νόμο, είτε από την παράδοση. Αλλά δεν υπάρχει κάποιο κοινοβούλιο που από μόνο το αυθόρμητο αποφασίζει να αλλάξει την έδρα όπου γίνονται οι σύνοδοι. Από όλα αυτά λοιπόν απορρέει, πρέπει να μάλλον τα λάβει κανείς όλα αυτά υπόψη για να σκεφτεί τη δυνατότητα να αλλάξει η έδρα του Ευρωκοινοβουλίου. Και εδώ μια διευκρίνηση. Πρέπει να διακρίνουμε, και αυτό δεν γίνεται πάντοτε στα έγγραφα που ασχολούνται με αυτό το θέμα, την έδρα από το χώρο εργασίας. Η έδρα ορίζεται ως το Στρασβούργο, όμως υπάρχουν άλλοι χώροι εργασίας, μέρη εργασίας, ε, τόποι εργασίας, όπως που είναι η Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο, οπουδήποτε αλλού. Το θέμα της τροποποίησης της έδρας λοιπόν είναι πολύ συγκεκριμένο, διότι αυτό ορίζεται από τη συνθήκη και για να αλλάξει η έδρα πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση των συνθήκων που θα πρέπει να γίνει μέσω της ελευθερία διαδικασίας που προβλέπεται από το άρθρο 48. Και εδώ η συμφωνία του, του 10 είναι πολύ σαφής και έχει αποφασιστεί, έχει μάλλον αναφερθεί σε διάφορες αποφάσεις. Είναι 97 και 2 της αποφάσης το 2012 κοινοβου... ότι τα κράτη μπορούν να αποφασίσουν πού είναι η έδρα του Ευρωκοινοβουλίου και ότι αυτό δεν εμποδίζει την εσωτερική ε, οργάνωση του Κοινοβουλίου αλλά φυσικά αυτή η δικονομία μπορεί να ξεπεραστεί από την αναθεώρηση του, των συνθήκων. Τα τρία λεπτά που μου απομένουν θα ήθελα να αναφέρω την διαδικασία και την κατάσταση άλλων κοινοβουλίων γιατί πιστεύω πως είναι χρήσιμο να κάνει κανείς μια σύγκριση και ξέρω πως ο συνάδελφος ε, εδώ έχει κάνει ε, έρευνες για αυτά τα θέματα. Καταρχήν, παραδείγματα εντός της Ένωσης. Αν δούμε το παράδειγμα της Πορτογαλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου ή τη Γαλλία, βλέπουμε ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσει το θέμα τη έδρα ε, δεν είναι απόλυτα υπό λοιπόν, τον έλεγχο του ίδιου του σώματος. Ε, εξαρτάται είτε από, την, από το Σύνταγμα, όπως στη Γερμανία, είτε από κάποιον νόμο, αλλά πάντως εν γέννη ένα κοινοβούλιο το ίδιο δεν μπορεί να τροποποιήσει το, την έδρα του ακόμα και σε περιπτώσεις όπου το σύστημα είναι άνω και κάτω βουλή. Το εκτελεστικό επίση εν γέννη δεν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει σε αυτή την υπόθεση. Αν δούμε τώρα καθεστώτα εκτό τη Ένωση, και εδώ ίσω ο παραλυσμό να είναι πιο σκόπιμο, διότι το πολιτικό σύστημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο κοντά στο αμερικανικό ή στο βραζιλιάνικο σύστημα. Στην περίπτωση της Βραζιλίας, ας πούμε, υπάρχει το σύνταγμα που λέει ότι η Ομοσπονδιακή Πρωτεύουσα είναι η Βραζίλια και ότι το, ε, το Κογκρέσο συνεδριάζει εκεί. Απλώ προβλέπεται ότι δεν υπάρχει σημαντικό λόγο. Η πλειοψηφία των βουλευτών μπορεί να αποφασίσει να συνεδριάσει σε άλλο τόπο, αλλά αυτό δεν έχει πραγματικά νόημα. Στη ε, ΣΥΠΑ είναι συγκρίσιμη κατάσταση. Το Σύνταγμα λέει πως όλα οι θεσμοί βρίσκονται στην περιοχή της Κολόμπια, μπορεί να αλλάξει μέσω του συντάγματος, αλλά το ίδιο το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ωστόσο, ε, σύμφωνα με το έθιμο, το Κογκρέσο συνεδριάζει εκεί που βρίσκονται οι, ε, οι συνεδροί του. Και άρα ε, ε, μπορούν, θα μπορούσε να συνεδριάσει και αλλού. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να γίνει κάτι τέτοιο. Αν δούμε τώρα την Ελβετία που έχουμε κοινό νομικό σύστημα και εκεί ε, ε, το κοινοβούλιο είναι πολύ αυτόνομο στην ιστορική του διοργάνωση, αλλά αυτό δεν περιλαμβάνει την επιλογή της έδρας του. Ωστόσο έχουν υπάρξει συνεδριάσεις στο Λουγκάνο, στη Γενέβη, στην ιστορία του Ελβετικού Κοινοβουλίου. Τώρα, το Παρλασούρ είναι μια περίεργη περίπτωση. Είναι το κοινοβούλιο του Μέρκοσούρ. Έχει γίνει πολλή λόγο για την έδρα αυτού του θεσμού και τελικά αποφασίστηκε να δημιουργηθεί αυτό το κοινοβούλιο και να εδρεύει εκεί όπου εδρεύουν και τα άλλα θεσμικά όργανα του Μερκοσούρ, δηλαδή στο Μοντεβιδέο. Ε, ενώ υπήρχαν εντάσεις ανάμεσα στις χώρες ώστε να γίνει κάποια κατανομή των εδρών των διαφόρων θεσμών στις διάφορες πόλεις και στις διάφορες χώρες. Να αναφέρω επίσης δύο περιπτώσεις κοινοβουλίων όπου το κοινοβούλιο δεν εδρεύει στην πρωτεύουσα. Στην πρωτεύουσα. Το κοινοβούλιο εδρεύει στο Σαντιάγκο. Ε, ε, στο Βαλπαραΐσο, ενώ η έδρα της κυβέρνησης είναι στο Σαντιάγκο. Ε, ε, γίνεται μια συζήτηση όμως τώρα για την επιστροφή του Κοινοβουλίου στο Σαντιάγκο. Και έπειτα Νότιος Αφρική συχνά αναφέρεται ως παράδειγμα. Υπήρχαν εντάσεις ανάμεσα στις τέσσερις επαρχίες για να πετύχουν την παρουσία πολιτικών θεσμών. Ε, αποφασίστηκε λοιπόν να συνεδριάζει στο Cape Town το Κοινοβούλιο, η κυβέρνηση στην Πρετόρια και το δικαστήριο σε μια άλλη πόλη. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει επιστημονική απάντηση στην αυτονομία, για την αυτονομία του Κοινοβουλίου. Δεν υπάρχει τίποτα στι θεωρίε που να λέει το απριορίο ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να έχει το, δικαίωμα να αποφασίζει για την έδρα του. Και δεν υπάρχει ούτε και κάποιο συστηματικό δικαίωμα των Κοινοβουλίων να αποφασίζουν για την έδρα του. Μάλιστα, μάλλον εξαίρεση είναι αυτό. Θα έλεγα λοιπόν ότι η απάντηση για το θέμα τη έδρα μπορεί να είναι μόνο πολιτική φύση ή διπλωματική φύση. Διότι το πολιτικό σύστημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει συγκεκριμένο ορισμό για το βαθμό αυτονομίας το οποίο μπορεί να χαίρει το Ευρωκοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη για την έλλειψη χρόνου ε, και την πίεση. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας συστήσω τώρα το δεύτερο μιλητή μας, το Ρίτσαρτ Βουέτεκερ, ε, που ε, είναι ελέκτρος στο Πανεπιστήμιο του Λάγκαστερ, ε, ε, του Λέστερ, συγγνώμη. Έχει κάνει ιδιαίτερη έρευνα για εθνικά κόμματα, για τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Έχει εργαστεί και για άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομοθεσία και συγκριτική λειτουργία. Έχει ε, συγγράψει διάφορα άρθρα και βιβλία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την συγκριτική πολιτική και πιο πρόσφατα οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η επιρροή των εθνικών κομμάτων και ε, νομοθετική εξουσία. Ε, στο Λονδίνο δημοσιεύτηκε αυτό το 2011 και με τον Σάιμον Χίξ έχει κάνει πολλές έρευνες μεταξύ ευρωβουλευτών για την εσωτερική οργάνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον καθορισμό των εδρών, πολλές και οι δημοσιεύσεις του ε, για την επιρροή των εθνικών κομμάτων ε, στις ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές του Κοινοβουλίου και γενικότερα στον 21ο αιώνα πώς λειτουργούν και πώς επηρεάζουν το σύστημα των επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα εθνικά κόμματα. Διάφορα λοιπόν ε, άρθρα και συγγράμματα αναφέρεται αυτό. Από το 1979 μέχρι το 1999 έχει μελετήσει μια 20 ετία ε, σε αυτά τα θέματα. Ε, Χαίρομαστε πάρα πολύ που βρίσκεστε ενώπιόν μας. Ήθελα να τα διαβάσω όλα αυτά για να σας συστήσω γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποιος είστε. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε να μιλήσω. Σε ένα θέμα που έχετε τόσα πολλά και σημαντικά ενδιαφέροντα, στην Επιτροπή δηλαδή που έχετε τόσα πολλά και σημαντικά, και σημαντικά ενδιαφέροντα θέματα. Μου ζητήσατε να μιλήσω για το δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτοοργάνωση. Να μπορεί κανεί να λάβει την απόφαση για το πώ οργανώνει την εργασία του, αυτό έχει και επιπτώσει ό,τι αφορά τη λογοδοσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέναντι στου ψηφοφόρου του. Επίση, αποτελεσματικότητα τη νομοθετική διαδικασία. Θα βασιστώ λοιπόν σε κάποιε πανεπιστημιακέ έρευνε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλα θέσει σχετικά θεσμικό όργανα. Πρώτα να μιλήσω για την κίνηση εντό και εκτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή από και προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τι σημαίνει αυτή η τάση σε ό,τι αφορά ένα πιο θεσμοποιημένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα φυσικό βήμα από το, την ελευθερία που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπω είπε και ο προηγούμενο μου, θα ήταν το Κοινοβούλιο να μπορεί να αποφασίζει πού έχει την εργασία του. Μιλώ επίση και για την ασυνήθη φύση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θεωρείται τμήμα ενό ε, ε, νομοθετικού οργάνου δύο σωμάτων που είναι λίγο δύσκολο να βρίσκονται διαφορετικέ πόλει. Μιλώ και για τι ε, ευνοϊκέ επιπτώσει που θα έχει η απόφαση του ίδιου του Κοινοβουλίου για το που θα τοποθετήσει τη θέση εργασία. του. Θα μιλήσω και για τι απόψει των Ευρωβουλευτών και θα τελειώσω σχετικά με το είναι ο τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να είναι υπόλογοι οι ευρωβουλευτέ για τι αποφάσει που λαμβάνουν για το πώ εργάζεται το Κοινοβούλιο. Από αυτά που γνωρίζουμε τώρα για την κίνηση προ και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το σύστημα επιτροπών του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φαίνεται να γίνεται σιγά σιγά πιο επαγγελματικό. Και να χρησιμοποιήσω ε, έναν όρο τη ε, κοινωνιολογική επιστήμη είναι πιο institutionalized, δηλαδή είναι πιο θεσμοποιημένο. Θα μπορούσε ο, ο να, μιλάει, να διαβάζει λίγο πιο αργά. Παρακαλούν πολύ διερμηνεί. Επίση, υπάρχουν και κάποια όρια μεταξύ των ε, ε, διαφόρων εδρών. Τώρα, μετά από τις ε, εκλογές του 1994, αυτό, αυτή η κίνηση των ευρωβουλευτών από 58% έχει πέσει κάτω από το 50% το 2009 και μετά. Είναι σχετικά υψηλή. Ακόμα πάντως είναι πτωτική η τάση. Αν εξετάσουμε τις αδειοδρομίες των ευρωβουλευτών από το 79 μέχρι το 99 πάνω από 36 από αυτού επανήλθαν ξανά και ξανά. Επομένω, ορισμένοι έχουν κάνει σταδιοδρομίες και έχουν μείνει παραπάνω από μία θητεία. Περισσότεροι ευρωβουλευτέ παραμένουν μάλιστα από μία θητεία σε άλλη στι ίδιε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ. Για παράδειγμα, πριν από τι προηγούμενε εκλογέ, μία από, τις, μία από πέντε έδρε παρέμειναν. Σε ό,τι αφορά τώρα του κατόχου των εδρών, αυτοί που έμειναν, ο αριθμό δηλαδή που έμεινε στην ίδια έδραση η Κοινοβουλευτική Επιτροπή αυξάνει σταθερά από χαμηλό σημείο το 94 πάνω από το 50% στις εκλογές του 2009. Επίσης για το ποιος λαμβάνει τις ηγετικές θέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνει ότι αυτοί που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία, μεγαλύτερη πείρα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνονται μάλλον αυτοί ε, πρόεδροι ε, ομάδων ή ε, διαφόρων άλλων σωμάτων. Τέτοιε αλλαγές αναμένει λοιπόν να δει κανεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εάν το Κοινοβούλιο πρόκειται να γίνει πιο θεσμοποιημένο, institutionalized δηλαδή, και επομένω να αυξήσει την νομοθετική του ε, επιρροή. Για να συνεχιστεί αυτή η εξέλιξη, το Κοινοβούλιο θα υποφεληθεί εάν μπορεί να αποφασίζει αυτό το που διεξάγει τι δραστηριότητέ του. Αυτό θα του δώσει και κάποιο, κάποια ευελιξία σχετικά με το χρονοδιάγραμμά του, που δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή. Τέτοια ευελιξία θα επιτρέψει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ανταποκρίνεται καλύτερα στα γεγονότα και να μοιράζει καλύτερα το φόρτο εργασία του. Η ελευθερία που απολαμβάνει τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπω είπε και ο φίλο μου Κώστα, του έχει επιτρέψει να αυξήσει τι εξουσίε του με τρόπο που δεν καλύπτονται από τη συνθήκη. Έχει de facto εξουσία λοιπόν ε, για να τροποποιήσει την ε, σύνθεση τη Κομισιόν που δεν περιλαμβάνεται στις συνθήκες. Από τότε όμως που ανέλαβε ε, η Επιτροπή Μπαρόσο έχει σημειωθεί αυτή η εξέλιξη στο Κοινοβούλιο. Επομένως το Κοινοβούλιο έχει την, ικανότη, έχει την εξουσία μάλλον να ρυθμίζει τα του κανονισμού του. Και επειδή έχει αυξηθεί και ο ρόλο του ε, θεσμικά, αυτό το ωφελεί. Το, αυτό που θέλω να πω τώρα είναι ότι το Κοινοβούλιο πολλοί πολιτιολόγοι το θεωρούν ως ένα ε, νομοθετικό όργανο από δύο, άνω και κάτω βουλή δηλαδή, που δεν μπαίνει όμως σε κανένα εθνικό πολιτικό σύστημα. Εδώ έχουμε το Συμβούλιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βέβαια, οι εξουσίες ε, ποικίλουν ανατομέα πολιτικής των οργάνων αυτών. Τώρα, να υπάρχει ένα κτίριο για, το ένα, για τη μία βουλή και άλλο κτίριο σε άλλη πόλη για άλλη βουλή, αυτό είναι ασύνηθες. Συνήθως μοιράζονται το ίδιο κτίριο και εάν όχι τουλάχιστον βρίσκονται στην ίδια πόλη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν και ως αποτέλεσμα των όσων περίγραψε ο καθηγητής κ. Κώστα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τροποποιηθεί από ό,τι ήταν στην αρχή. Έχουμε λοιπόν μια πολύ διαφορετική οργάνωση από την αρχή όταν είχαν προσωρινά καθοριστεί στα 1950 οι έδρε των θεσμικών οργάνων. Δεν χρειάζεται βέβαια να σα το πω εγώ ότι η διάδραση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου των Υπουργών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η βάση για την νομοθεσία με τις διάφορες διαδικασίες, τη συνήθως νομοθετική διαδικασία ή τον τριμερή διάλογο. Και αν τώρα η έδρα του Κοινοβουλίου έχει κάποιο ρόλο να παίξει στην αποτελεσματικότητα, αυτό, είναι αυτό είναι, σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να μπορεί να τα ε, αποφασίζει. Ως γνωρίζουμε από τις, ε, ε, ε, έρευνες που έχει κάνει η ομάδα ερευνών του Κοινοβουλίου, 52% των βουλευτών έχουν πει ότι συναντώνται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα με ομάδες ε, συμφερόντων. Πάνω από το 1 πέμπτο έχουν πει ότι έχουν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα επαφές με προσωπικό τη Κομισιόν. Και πάνω από 70% τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Όλες λοιπόν αυτές οι συχνές επαφές δείχνουν επίση ότι το Κοινοβούλιο θα ωφεληθεί από το αν παραμείνει σε μία πόλη. Τώρα το να μπορέσει το Κοινοβούλιο να αποφασίσει μόνο του, αυτό θα του επιτρέψει και κάποια ευελιξία και στον καθορισμό του χρονοδιαγραμματό του. Κάτι που είναι σύνθεση για πολλά εθνικά κοινοβούλια. Για την ώρα, οι περισσότερε ψηφοφορίε γίνονται όλε μαζί σε ορισμένα χρονικά σημεία στι περιόδου συνόδου του Στρασβούργου. Δηλαδή δεν έρχονται αμέσω μετά τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος. Και το Jacobs Book και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνει ότι πολλοί ε, παρατηρητέ εκ των έξω το βρίσκουν αυτό πάρα πολύ πάρξενο. Για παράδειγμα το Βρετανικό Κοινοβούλιο συνήθως οι ψηφοφορίες γίνονται αμέσως μετά τη συζήτηση και σε πάνω από 70% με δίνοντας έτσι την ευκαιρία να παρακολουθούν αμέσως όσοι παρακολουθούν δηλαδή τη συζήτηση και μετά την ψηφοφορία. Είναι σύνηθες επίσης σε ορισμένα ε, νομοθετικά σώματα συνεδριάσεις επιτροπών ακροάσεις να γίνονται την ίδια μέρα μαζί με τις διαδικασίες, με τις ε, ε, συνόδους μάλλον ε, Τη Ολομέλεια. Αυτό θα προσφέρει επίση ε, την απαραίτητη ευελιξία στην οργάνωση του Κοινοβουλίου. Ένα άλλο θέμα είναι ότι ω προκύπτει από έρευνε, φαίνεται ότι μια πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών υποστηρίζουν την διεξαγωγή των Ολομελιών στι Βρυξέλλες. Το γνωρίζουμε αυτό από έρευνε, όπω είπα μεταξύ των Ευρωβουλευτών μεταξύ 2000 και 2006 και 2010 και βλέπουμε εν τέλει ότι περίπου 70% των Ευρωβουλευτών συμφωνούν ότι θα πρέπει το Κοινοβούλιο να μπορεί να διεξάγει όλες τις ολομέλειές του στις Βρυξέλλες. Τέλος, οι Ευρωβουλευτές αντιμετωπίζουν αρνητική κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τους λόγους αυτούς. Εάν είχαν λόγο οι ευρωβουλευτές για το πού θα οργανώνουν τις εργασίες τους, αυτό θα επέτρεπε και στους ε, ψηφοφόρους και επομένως και στα μίδια να τους θεωρούν πλέον υπόλογους. Και αυτό βρίσκω ότι είναι σημαντικό επιχείρημα για να χορηγηθεί στο Κοινοβούλιο το δικαίωμα να αποφασίζει πού εντοπίζει την εργασία. Ε, Ευχαριστώ πολύ ε, και για την τήρηση του χρόνου και το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό. Πριν δώσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή, θα ήθελα να γνωρίσω πόσοι αγαπητοί συνάδελφοι θέλουν να μιλήσουν για να μοιράσουμε το χρόνο δίκαια. Βεβαίως και οι συγκητές αλίμονο. Λοιπόν, παρακαλώ να δηλώνετε για να σημειώνουμε τα ονόματά σας. Σηκώστε τα χέρια σας για να σας δούμε και να σας σημειώσουμε. Uh, ναι, ναι, κύριε Ροζέλη, είστε πρώτος έτσι κι αλλιώς ε, στο κατάλογο. Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών γιατί μπορεί να έρθουν και άλλοι συνάδελφοι, αλλά να γνωρίζω πάνω κάτω πόσοι θα είναι οι συνάδελφοι που θα πάρουν το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα ήθελα να δώσω ε, το λόγο στον κύριο Χέρβικ Χόφμαν που είναι καθηγητής Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου. Ένα μικρό βιογραφικό του, όπως σας είπα είναι καθηγητής ε, στην έδρα Ζαμονέ, Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου. Ήταν επισκέπτη στο Σιαν Πο στο Παρίσι, στο Κολόμπια Νομική και Ινστιτούτο Δημόσια Διοίκησης. Στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου ίδρυσε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Δικαίου. Ω μέλος του Δικηγορικού ε, Συλλόγου της Κολονίας ε, μπορεί ε, να αγορεύει ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Επίσης έχει δημοσιεύσει μεγάλο έργο για το διοικητικό δίκαιο στην Ευρώπη. Ε, συμμετέχει ε, σε διάφορα περιοδικά και είναι ιδρυτικό μέλος ε, του ερευνητικού δικτύου για το Ευρωπαϊκό Διοικητικό Δίκαιο και το Ευρωπαϊκού Δικαίου. Και επίσης γερμανικά έχει δημοσιεύσει για την ε, ιεράρχη ε, των κανόνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο και γενικότερα για διάφορα ευρωπαϊκά θέματα και διοικητικά. Είναι πάρα πολύ πλούσιο και το βιογραφικό του όσο και το έργο του. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε τόσο καταπληκτικούς και αξιόλογους ε, σήμερα εκπροσώπους και εμπειρογνώμες. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. συνεχίζω από εκεί που σταμάτησα οι προλήσατες και θα μιλήσω για τρία θέματα. Πρώτον, το υπόβαθρο, την αρχή. Δεύτερο, πώς θα μπορέσει κανείς να το ε, χειριστεί και να το ε, εξελίξει. Ε, τα τελευταία 60 χρόνια ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε αναπτυχθεί με τρόπο διαφορετικό από τα άλλα θεσμικά όργανα και με απόλυτους όρους αλλά και με σχετικούς όρους. Ε, στον προϋπολογισμό, στα νομοθετικά έχει κερδίσει εξουσίες και ε, επίσης είναι υπόλογη εκτελεστική εξουσία και μπορεί να την καλέσει το Κοινοβούλιο να βοηθεί, αλλά όπως γνωρίζουμε δεν μπορεί να αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κυρίαρχα για τους τόπους εργασίας και την έδρα. Αν δούμε τα 27 και προσεχώ 28 κρατη έξι τουλάχιστον, έχουν ε, διάταξη και πρόβλεψη στο Σύνταγμά τους που ορίζει την έδρα του Κοινοβουλίου τους. Δανία, Ιρλανδία, Λετωνία, Λουξεμβούργο, Σουηδία. Ωστόσο, αν έρθετε να μελετήσετε τις διατάξεις, ε, βλέπετε ότι εδρεύει στην ίδια πόλη η ε, νομοθετική με την εκτελεστική εξουσία. Ενώ οι λεπτομέρειες στις ευρωπαϊκές συνθήκες ε, κατά πολύ υπερβαίνουν τις εθνικές ρυθμίσεις. Λοιπόν, ποια είναι αυτή η αυτοοργάνωση. Είναι η εξουσία αλλά και η υποχρέωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αυτοοργανώνεται όπως αναφέρεται ε, τη συνθήκη και το άρθρο 232, συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τον εσωτερικό του κανονισμό. Και αυτό έχει ερμηνευτεί σε διάφορες αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων λέγοντας ότι θα πρέπει να λαμβάνει απαραίτητα μέτρα για να διεξάγεται σωστά η λειτουργία του κοινοβουλευτική. Είναι υποχρεωμένο λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από αυτού του όρου να αυτοοργανωθεί. Ε, δηλαδή να δώσει ε, ένα περιεχόμενο στις πρόνοιες της συνθήκης. Καλείται λοιπόν το Κοινοβούλιο να αυτοοργανωθεί με βάση τις εξουσίες που του δίδει η συνθήκη. Τώρα, Αν δούμε το πλαίσιο αυτού του δικαιώματο του Κοινοβουλίου στην αυτοοργάνωση, και πολύ γρήγορα ερχόμαστε στο άρθρο 341 και το πρωτόκολλο υπαριθμών 6, μιλώντας για την έδρα. Το άρθρο 341 της Συνθήκης για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι με κοινή συμφωνία των κυβερνήσεων των, των μελών ε, ορίζεται η έδρα των θεσμικών οργάνων. Είναι περίεργη αυτή η ε, ρύθμιση και όπως γνωρίζετε η απόφαση του Δημιουργού στη συνέχεια έγινε πρωτόκολλο 6 ε, στην συνθήκη του Άμστερνταμ και στις επόμενες συνθήκες που ακολούθησαν που είναι πρωτογενές δίκαιο η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι το πλαίσιο που ισχύει το νομοθετικό. Τι μπορεί να κάνει τώρα το Κοινοβούλιο αν φρονεί ότι είναι απαραίτητο κάτι να αλλάξει σε αυτό το πλαίσιο. Ιδιαίτερα σε σχέση με την έδρα του. Δύο είναι οι προφανείς δυνατότητες. Το ένα είναι η τροποποίηση των συνθηκών και το άλλο να ε, διερευνηθούν τα όρια της παρούσας ε, κείμενης συνθήκης. Έρχομαι στην τροποποίηση τώρα των συνθηκών. Τρεις είναι οι δυνατότητες. Πρώτον, να διαγραφεί το, άρθ, το πρωτόκολλο 6. Αυτό θα ήταν ε, κακή ιδέα γιατί θα παραμείνει ενισχύει το άρθρο 341 της συνθήκης που οδήγησε και στην απόφαση του Εδιμβούργου η οποία θα εξακολουθεί να ισχύει ακόμα και αν καταργηθεί το πρωτόκολλο υπ. 6. Η δεύτερη δυνατότητα είναι να διαγραφούν και τα δύο, και το άρθρο 341 και το πρωτόκολλο 6 και αυτό τι θα σημάνει στην πράξη ότι το δικαίωμα αυτοργάνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματο να ορίζει την έδρα του και του τόπου εργασίας, παράδειγμα μέσω του κανονισμού του εσωτερικού για τη λειτουργία του, ε, θα συνεχίσει να ισχύει. Ωστόσο, αυτό το δικαίωμα θα πρέπει να ασκείται υπό την υποχρέωση ειλικρινού συνεργασία με τα αντίστοιχα κράτη-μέλη. Ωραία, αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία ελευθερίας κινήσεων ε, και μπορεί, επίσης το τρίτο είναι να τροποποιηθεί το άρθρο 341 και το πρωτόκολλο 6. Με λεπτομέρειες που θα αποφασιστούν και κατά τα άλλα και το ΔΕΚ δεν έχει δικαίωμα να αναθεωρήσει το περιεχόμενο του πρωτογενούς δικαίου, μόνο τις διαδικασίες που οδηγούν στην ε, αναθεώρησή του. Ε, Δηλαδή μπορεί να επανακαθοριστεί η έδρα ενδεχομένως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έτσι ή να οριστεί ε, ο τρόπος, η ε, τόπη εργασίας. Για να αναθεωρηθεί η συνθήκη χρειάζεται κύρωση από όλα τα κράτη-μέλη, αλλά προηγουμένως κάνει πρόταση το Κοινοβούλιο εφόσον το επιθυμεί και μπορεί να το πράξει σε ε, μια συμφωνία δέσμη, ας πούμε, για περαιτέρω διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα πλαίσια άλλων προτάσεων που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, όπως έχει ανακοινώσει εξαγγείλει. ανακοινωσει εξαγγειλη πρόταση μπορούν να κάνουν όλα τα θεσμικά όργανα στο Συμβούλιο, που το αποστέλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει αν χρειάζεται να ε, συγκληθεί συντακτική συνέλευση ή όχι. Αλλά και η διακυβερνητική διάσκεψη, και αυτό έχει σημασία, ε, με κοινή συμφωνία, βλέπε ομοφωνία, ορίζει ποιε θα είναι οι τροποποιήσει που θα γίνουν στι συνθήκε και μετά χρειάζεται να κυρωθεί η συνθήκη. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη βεβαίω που ενδεχομένω να αντιδρούν στην αλλαγή ε, τη επίσημη έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βέβαια, οποιαδήποτε διαδικασία τροποποίηση αναθεώρηση των συνθηκών έχει και κινδύνου. Δηλαδή, μπορεί στι διαπραγματεύσει, τα πράγματα να προκύψουν διαφορετικά από εκείνα που θα επιθυμούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου ε, μπορεί να ξανανοίξει όλο το θέμα των εδρών, ιδιαίτερα για τις χώρες που μπήκαν μετά το 2004 και δεν έχουν τόσους πολλούς οργανισμούς, θεσμικά όργανα, ε, να θέλουν να αυξηθεί το μερίδιό τους. Καλά, αυτό απομένει να φανεί. Αυτές είναι οι δυνατότητες. Υπάρχουν εναλλακτικέ όμως ως προς την αναθεώρηση των συνθηκών. Και το ερώτημα προφανώς είναι ε, τι περιθώριο ε, ε, χειρισμών έχει το Κοινοβούλιο στην κείμενη νομοθεσία. Και αυτή είναι η νομολογία του ΔΕΚ, ιδιαίτερα το 1997 και το 2012. Έρχεται εδώ να επηρεάσει. Και ποια είναι τα βασικά ο ακρογωνιαίος λήθος, ότι ασκώντας το δικαίωμα αυτοοργάνωσης του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να σέβεται τις αρμοδιότητες και εξουσίες των κρατών μελών να ορίζουν την έδρα του. Να ορίζουν την έδρα του. Αλλά το πρωτόκολλο υπαριθμών 6 θα πρέπει να ερμηνεύεται ε, με τρόπο ώστε να θεωρεί τη βασική έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Στρασβούργο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει από εκεί και πέρα το Κοινοβούλιο την ευχαίρεια να ορίζει τη λειτουργία του και τι εσωτερικέ κοινοβουλευτικέ εργασίες. Ναι, βέβαια Σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι ορισμένες αλλαγές στον τρόπο εργασίας του Κοινοβουλίου είναι θεμητές. Ήδη το χρονοδιάγραμμα έχει τροποποιηθεί και υπάρχει και αντίστοιχη νομολογία του δικαστηρίου και έχουμε και πολύ ε, σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα υπάρχουν αυτές οι αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα. Υπάρχουν 12 τακτικές σύνοδοι που πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται στο Στρασβούργο και κάποιες έκτακτες. Ε, βέβαια, η σημαντικότερη είναι η σύνοδο Ολομέλεια για τον προπολογισμό και ορίζεται και ρητά, αλλά δεν υπάρχει σαφής ε, ρύθμιση για το ποια θα είναι η διάρκεια. Δεν πρέπει να είναι απαραίτητο μία εβδομάδα. Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες που μπορούν να διερευνηθούν. Θα μπορούσαμε να μπούμε σε λεπτομέρειες τώρα. Δεν έχω το χρόνο, αλλά με χαρά να το συζητήσουμε αν το επιθυμείτε. Υπάρχουν ε, προφανώς δυνατότητες να εργαστεί κανείς εντός του πλαισίου του εφισταμένου δικαίου για να βελτιωθεί η λειτουργία του Κοινοβουλίου και να σταματήσει αυτός ο πλανόδιος θίασος, αυτό το τσίρκο όπως κοινώ το γνωρίζει ο κόσμος. Γίνονται διάφορες συζητήσεις, ε, βέβαια για τα τεχνικά ζητήματα εσείς είστε πιο ε, από μένα, αλλά ε, πριν τελειώσει ο χρόνος μου θα ήθελα να πω το εξής. Ε, στα πλαίσια του δικαιώματο αυτοοργάνωση έχει το Κοινοβούλιο το δικαίωμα να προβεί σε συμφωνίες με τα κράτη-μέλη. Το έχει πράξει ήδη με το Λουξεμβούργο, όπου συμφώνησε το Λουξεμβούργο 50% του προσωπικού να εδρεύει μόνο στο Λουξεμβούργο αντί το σύνολο του προσωπικού και αυτό είναι ε, σε αντίθεση με τα όσα ορίζουν οι συνθήκες, θα μπορούσαν να βρεθούν και λύσεις για το Στρασβούργο μετά από συνεννόηση με τη Γαλλία για να γίνει πιο εύκολη η λειτουργία τουλάχιστον μέχρι να τροποποιηθεί ε, η συνθήκη. Συμπεραίνω λοιπόν σύντομα πλήρης αναθεώρηση της συνθήκης θα μπορούσε να ρυθμίσει το θέμα της έδρας, αλλά υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, μπορεί να είναι και απαραίτητο να ε, δοθεί έτσι μια λύση ριζική και καθαρή, αλλά υπάρχουν ακόμα και δυνατότητες βάσει βάση την κείμενη νομοθεσία να διερευνηθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Χρειάζεται αλλαγή των συνθήκων. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι <laughs> διευρύνεται όσο πάει η εικόνα μας. Επόμενος συνάδελφος είναι από τη Γερμανία ο Ανδρέας Μάουρερ, Διευθυντής του Γερμανικού Ινστιτούτου ε, Θεμάτων Διεθνών και ε, Θεμάτων Ασφαλείας της Βρυξέλλης. Είναι επίσης καθηγητής πολιτικών επιστημών και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στο Πανεπιστήμιο του Ινσπρουκ. Είναι μέλος του ε, Συμβουλευτικού Συμβουλίου του Παρατηρητηρίου Κοινοβουλίων μετά τη Συνθήκη Λισαβόνας έχει εργαστεί ως Εθνικός Εμπειρογνώμων στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Κοινοβουλίου ε, και ήταν επίσης ε, σύμβουλος στην ε, Ευρωπαϊκή Συντακτική Συνέλευση με ευρύ έργο και δημοσιεύσεις για τα κοινοβούλια και τον κοινοβουλευτισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαπραγματεύσεις για τη μεταρρύθμιση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναθεώρηση των συνθήκων. Τα περισσότερα δημοσιεύματα, η του είναι στα γερμανικά, να μην σας τα διαβάσω. Αν θέλετε μπορώ ε, απλώς ήθελα να σας πω ότι δεν έχω πρόβλημα, μπορώ και να τα διαβάσω. Ε, ε μία από τις δημοσιεύσεις είναι στα αγγλικά. Ε, το έχετε στους φακέλους σας. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ. Thank you, Chair. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Όταν με προσκαλέσατε να μιλήσω για το θέμα αυτό, προσπάθησα να προβώ σε μία διάκριση αυτού του δικαίου αυτοοργάνωσης που θα έλεγε self-organization στα αγγλικά, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Το ένα είναι το δικαίωμα αυτοδιοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ε, υλοποιείται μέσω του κανονισμού των αποφάσεων του Προεδρείου του συνηθισμένων αποφάσεων των Επιτροπών, διαθεσμικών συμφωνιών, δηλαδή διάφορες αποφάσεις και άλλα που επιτρέπουν την καλύτερη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Και κυρίως για να διαμορφώνονται οι διαθεσμικές διαδικασίες βασισμένες στην αποτελεσματικότητα της συνεργασίας, επατελεσματικότητα της διαδικασίας και του πολιτικού κύκλου. Υπάρχουν και άλλα επιχειρήματα που προβάλλονται υπέρ της συγκέντρωσης της διαδικασίας αυτής στις ίδιες τις Βρυξέλλες. Υπάρχει δηλαδή και το περιβαλλοντικό επιχείρημα με την αποφυγή των ταξιδιών στο Στρασβούργο, το, της δημόσιας εικόνας του οργάνου, οι, εργασίες, ε, οι συνθήκες εργασίας ε, βουλευτών και προσωπικού, τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζονται, οι ακαταλήμματα στο Στρασβούργο κλπ. Αυτή είναι μια πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά που έχει σχέση βέβαια με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηριού, με τα επιχειρήματα που έχουν προβάλει ορισμένες ε, σημαντικές χώρες μέλη. Εκεί βεβαίως παίζει ένα ρόλο και η αυτοδιάθεση του θεσμικού οργάνου. Το δικαίωμα δε των χωρών μελών να καθορίζουν που ε, μέσω του άρθρου 341 τώρα της ε, συνθήκης που λέει ότι συμφωνούν οι χώρε μέλη, ούτε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ούτε Συμβουλίο Υπουργών, ούτε τίποτα. Και αυτό ε, μπαίνει και στο παράρτημα υπαριθμών 6. Εκεί λέει αυτοδιάθεση των χωρών μελών ω αφεντικών της συνθήκη, ω κυρίων της συνθήκη. Όλα εξαρτώνται από τι χώρες μέλη που είναι οι πατέρε και μητέρες της ε, συνθήκης και της Ένωσης. Η άσκηση αυτού του δικαιώματο περιλαμβάνει και τον καθορισμό τη έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και του είδους των δραστηριοτήτων που θα ε, διεξάγονται εκεί. Και αυτό τα λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τώρα από την άλλη μεριά το επιχείρημα που ε, προβάλλεται υπέρ της συγκέντρωσης των εργασιών του Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες το 2006 και το 2010 εκφράστηκαν τα μέλη του δεν άλλαξε πολύ η άποψή τους αυτή το 2010, 70 περίπου τις 100 των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που απάντησαν τουλάχιστον στο ερωτηματολόγιο λένε ναι είμαστε σαφώς υπέρ να μπορούμε να διεξάγουμε όλες τις ολομέλειές μας στο Στρασβούργο. Να μας το επιτρέψουν δεν σημαίνει κιόλας ότι θα το κάνουμε αλλά θέλουμε να έχουμε τουλάχιστον τη δυνατότητα να μπορούμε να το πράξουμε εφόσον το επιθυμούμε. Να και μια σύγκριση εδώ σε άλλες χώρες μέλη, όχι τρίτες χώρες, Εγώ βρήκα παραλλαγές μεταξύ τριών δυνατοτήτων. Αφενός διεθνείς οργανισμοί ή συντάγματα που προβλέπουν την πρωτεύουσα ε, μιας χώρας, εδώ βεβαίως ε, ε, ιδίως η Γαλλία, η οποία βέβαια τάσεται υπέρ του Στρασβούργου, μετά διεθνώς η οποια βεβαια τάσσεται υπερ του στρασβουργου μετα διεθνως η αργεντινη για διεθνείς οργανισμούς, οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ο ΑΣΕ, το ΝΑΤΟ κτλ. Δεν λένε τίποτα για έδρες. Στην άλλη πλευρά του φάσματος υπάρχουν ορισμένες η δηλαδή των χωρών μελών που λένε κάτι για την έδρα όπως Αυστρία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Σουηδία και διεθνώ η Νότια Αφρική είναι ενδιαφέρον το παράδειγμα αυτό, οι Ενωμένε Πολιτείε και διεθνεί οργανισμοί. Λίγο βέβαια ο χάρτη του ΑΣΕΑΝ που λέει καθαρά σε άθρο ότι κάθε χώρα μέλος του ΑΣΕΑΝ διορίζει μόνιμο αντιπρόσωπο στην Τζακάρτα. Δεν λέει ότι η πρωτεύουσα είναι η Τζακάρτα, αλλά κατ' εφαρμογή του άρθρου αυτού είναι προφανές ότι η Τζακάρτα είναι η έδρα. Τα παραδείγματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τώρα για περαιτέρω προβληματισμό μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ενδεχομένως για μια συνέλευση για να τροποποιηθεί η τρέχουσα κατάσταση Είδα λοιπόν τι κάνουν οι χώρες και βρήκα δύο παραδείγματα ενδιαφέροντα. Αφενός στην Ιρλανδία που λέει το Σύνταγμα καθορίζει ως έδρα του Προέδρου το Δουβλίνο ή κοντά στο Δουβλίνο. Και το Κοινοβουλίο επίσης λέει ε, καμιά φορά. Στη Σουηδία λέει λέει ότι ε, γίνονται στη Στοχόλμη αλλά και αλλού εφόσον το απαιτεί η ασφάλεια του σώματος. Η Αργεντινή διεθνώ λέει ότι ότι οι ε, κοινοβουλευτικές εργασίες οργανώνονται στην πρωτεύουσα η οποία καθορίζεται με νόμο του Κοινοβουλίου. Άρα δεν είναι δηλαδή σε ε, επίπεδο ε, συνταγματικού νόμου. και ούτω καθεξής. Αυτά τι σημαίνουν τώρα στην πράξη. Αν θεωρήσουμε δεδομένη, δεδομένο τον περιορισμό της αυτοδιάθεσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 341, δηλαδή δηλαδή καθήκον των χωρών μελών να καθορίζουν την έδρα των θεσμών, θα χρειαστεί λοιπόν να προσφύγουμε στο άρθρο 341 ή στο παράδειγμα 6. Δεύτερο, θα έπρεπε να γίνουν τροπολογίε από αυτόν. Με ποιο στόχο θα πρέπει να γίνει μια διάκριση, πρέπει να επαναπροσδιοριστούν οι έδρες και πού βρίσκονται οι έδρες αυτές. Θα πρέπει να αλλάξει η διατύπωση με κοινή συμφωνία των χωρών μελών ώστε να προσαρμοστεί στο 48 στο 48 μάλλον της συνθήκης ώστε να διευκολυνθεί η αλλαγή. ή προτιμάτε να αγωνιστείτε υπέρ της δημιουργίας του δικαιώματος αυτοδιάθεσης όπως η Νότια Αφρική, όπως η Αργεντινή που λένε ότι αποφασίζει το θεσμικό όργανο με παράγωγη νομοθεσία το που θα ε, εγκαταστήσει την έδρα του. Αυτές είναι οι δυνατότητες. Υπάρχει λοιπόν το 48, 6 ή 7 της απλουστευμένης διαδικασίας, εγώ μάλλον το αποκλείω αυτό, το 7 μάλλον όχι, διότι ε, είναι περιοριστικό των διαδικασιών στο Συμβούλιο Υπουργών, άρα δεν αποδίδει εν προκειμένου. Δεύτερη δυνατότητα, το 48 παράγραφος 3, απλοποιημένη ε, απλή ε, αναθεώρηση και εγώ το βρίσκω κάπως απίθανο διότι η έκταση τέτοιας αλλαγής θα σήμαινε περιορισμό των εξουσιών της Γαρίας και του Λουξεμβούργου και δεν θα το επιτρέψουν. Άρα η μόνη δυνατότητα που έχετε είναι η 48 παράγραφος 3 για το 2015 έχοντας υπόψη βέβαια ότι και τότε θα χρειαστεί ένα τεράστιο πακέτο δεν μπορεί να περιοριστείτε μονάχα στην έδρα και μέρος της δέσμης αυτής θα πρέπει να είναι και τι θα γίνει εφόσον οι Βρυξέλλες γίνουν έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πώς δηλαδή αντισταθμίζεται για τις απώλειες, ε, πώς αποθυσιμιώνεται δηλαδή το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο για τις απώλειες, τις ζημίες που θα έχουν. Το Ευρω... Ίσως το Λουξεμβούργο να γίνει European City of Justice και διαφορετικά. Μάλλον απίθανο ένας Γερμανός να ταχθεί υπέρ του Λουξεμβούργου ή της Γαλλίας, αλλά το θέμα αυτό, ότι θα έπρεπε να έχουμε περισσότερη αυτοδιάθεση για το πού θα είναι η έδρα μας, έχει σχέση με την αποτελεσματικότητα. Εγώ εργάστηκα για χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έκανα ταξίδια αυτά μεταξύ Βρυξελών και Στρασβούργου και δεν άλλαξε το αίσθημα που είχα ότι μια μεγάλη διαφορά μεταξύ Βρυξελών και Στρασβούργου είναι όταν το Κοινοβούλιο μετακινείται στο Στρασβουργό, μπαίνει σε ένα είδος διαρκού κονκλάβιου. Δηλαδή δεν υπάρχουν τόσα πολλά λόγια, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση έξωθεν. Αν θέλει λοιπόν το προσωπικό να, συναντήσει, ε, να συναντηθεί με ένα μέλο, με ένα βουλευτή για να συζητήσει τροπολογίε. ή αν το προσωπικό θέλει να συναντηθεί μεταξύ του για να καθίσει να βρει συμβαστικέ τροπολογίε κλπ. Εγώ τουλάχιστον είχα την αίσθηση αυτό δεν έχει καμία ε, πολιτική προέκταση, ότι είναι πολύ ευκολότερο να λειτουργήσουν τα πράγματα αυτά στο Στρασβούργο, όπου δεν υπάρχει όλο αυτό το πέρα δόθε, το μπες των μη κρατικών οργανισμών, των λόμπι, όπου το Κοινοβούλιο κάθεται και δουλεύει χωρίς όλα αυτά. Άρα να μην δούμε μονάχα τα της αυτοδιάθεσης, αλλά αν υπάρχουν και λόγοι να ταχθεί κανείς υπέρ τη έδρα αυτή του Στρασβούργου, τουλάχιστον για αυτέ τι τρει-τέσσερι μέρε, έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να μπορεί να λειτουργήσει ελεύθερο και ανεξάρτητο από του άλλου θεσμού, από τα άλλα θεσμικά όργανα. Σας ευχαριστώ. Θέλαμε να τονίσουμε μέσω αυτής της ακρόασης το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για το Ευρωκοινοβούλιο και για τα Εθνικά Κοινοβούλια, ιδιαίτερα όσον αφορά το δικαίωμα να οργανώνουν τις εργασίες τους και να δούμε πώς έτσι θα μπορούσε να αναπτυχθεί αυτό το δικαίωμα του Κοινοβουλίου στο μέλλον. Αφού έχουμε δύο συνεισηγητέ, όπω συμφωνήσαμε, ο πρώτα ο, κύριο, ο αντιπρόεδρος κύριος Φόξ θα πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ κυρίες και κύριοι και ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονές μας που ήρθαν στην σημερινή ακρόαση. Θα γνωρίζετε ότι η έκθεση την οποία συντάσσουμε εγώ και ο Κέραλτ αφορά την έδρα των Ευρω... τις έδρες μάλλον, των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Ε, έχουμε φτιάξει ένα έγγραφο εργασία και θα το βρείτε στο σημείο 6 των εγγράφων ε, τη Επιτροπή σήμερα και έχουμε αύριο μάλιστα συζήτηση για το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου εργασία. Γι' αυτό θα ήθελα να καλέσω σήμερα τα μέλη να υποφεληθούν ε, της παρουσίας των εμπειρογνωμόνων. Αν έχετε επικρίσεις ή για σχόλια για το έγγραφο εργασία μου, ας τα ακούσουμε αυτά αύριο. Σήμερα έχουμε μια κρόαση για το δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην διοργάνωση των εργασιών του και θα παραδεχτώ ότι ως Βρετανός συντηρητικός δεν είμαι από αυτούς που θέλουν να δώσουν περισσότερες αρμοδιότητες στο Ευρωκοινοβούλιο. Οι δικές μου ε, ανησυχίες είναι πρακτικής φύσης, πρακτικές με την έννοια ότι το πρωτόκολλο 6 λέει ότι θα έχουμε 12 συνόδους ολομελίας στο Στρασβούργο, θα έχουμε τις συνεδριάσεις των επιτροπών μας στις Βρυξέλλες. Και αυτό καταλήγει σε 200, εκατομμύρια ευρώ φορολογουμένων, των φορολογουμένων που σπαταλώνται λόγω των δύο εδρών πολλές ποσότητες, τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα, ενώ πηγαινορχόμαστε ανάμεσα στις γέδες, ενώ το Ευρωκοινοβούλιο διακηρύσει στον υπόλοιπο κόσμο πόσο σημαντική είναι η μείωση των εκπομπών. Και επίσης δαπανάτε ένα τεράστιο νούμερο χρόνου, ορών εργασίας των ε, υπαλλήλων μας, καθώς πηγαίνουν ανάμεσα στις γέδρες. Τώρα, Θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός όταν λέω ότι δεν, είμαστε, δεν, δεν εκφραζόμαστε στο κατά πόσο το, η η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διότι κατανοούμε απολύτω ότι κάθε κράτος έθνος έχει βέτο. Και γι' αυτό ε, δεν θέλουμε αυτό να αποτελέσει θέμα ανάμεσα στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο και το Λουξεμβούργο. Ακόμα και αν είναι απόφευκτο, όλοι θα γνωρίζουν τις πρακτικές συνέπειες όσον αφορά το, τις συνταγματικές αλλαγές. Εγώ η κατεύθυνση που θέλω να ακολουθήσει αυτή η έκθεση είναι μια αλλαγή στις ευρωπαϊκές συνθήκες που θα οδηγήσει στο να αποφασίσει το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο πού θα βρίσκεται η έδρα του. Και αυτό Μπορεί να είναι στη στο Στρασβούργο. Και εγώ θεωρώ ότι το Στρασβούργο πολύ πιο όμορφη πόλη από ότι οι Βρυξέλλες. Πολύ πιο ευχάριστο να εργάζεται κανείς στο Στρασβούργο και δεν είναι τόσο βρώμικη όσο οι Βρυξέλλες. Το Στρασβούργο είναι απείρως καλύτερη πόλη να εργάζεται κανείς. Όμως το θέμα είναι ω ε, αρχή, αν πρέπει το Συμβούλιο να αποφασίζει που θα συνεδριάζει το, το, το Κοινοβούλιο. Γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτή η ρύθμιση που ισχύει τώρα προκαλεί τεράστια ζημιά στη φινιστεροφημία του Κοινοβουλίου και στην Ένωση εν γέννη. Και θα έλεγα μάλιστα και στους τέσσερις εμπειρογνώμονες ότι σχεδόν σε κάθε συνεδρίαση, σε κάθε meeting στη δική μου περιφέρεια αυτός ο παραλογισμός αναφέρεται και θεωρείται ως λόγος να είναι κανείς κατά της ε, Ένωσης και να την επικρίνει γιατί λέει το ένα και κάνει το άλλο. Άρα λοιπόν το ερώτημα που θέλω εγώ να θέσω στους εμπειρογνώμονες μας όταν θα ολοκληρώσουν στο τέλος και ο κύριος Χόφμαν και ο κύριος Μάουερ το ανέφεραν ακροθυγώς είναι ποιο είναι ο πιο πρακτικός τρόπος όσον αφορά τροπολογία της συνθήκης, τροποποίηση της συνθήκης. Ποιο είναι ο πιο πρακτικός τρόπος για να επιτέχω αυτό που θέλω εγώ. Τροποποιώντα το 341, τροποποιώντα το πρωτόκολλο 6 και ίσως όταν θα ακούσετε και τα άλλα σχόλια των άλλων ευρωβουλευτών θα επανέλθετε και θα μου πείτε αυτό πρέπει να κάνετε. Να φτιάξετε έτσι το άρθρο 6 ή το 341 ώστε να λέει το τάδε. Γιατί στο τέλος της έκθεσης όταν θα με ψηφίσουμε για από αυτού στην Ολομέλεια, αυτό που θα ήθελα εγώ να βρίσκεται στο τελικό προϊόν, μια τροπολογία που σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο αποφασίζει πού συνεδριάζει. Αλλά δεν καταλήγουμε στο να διευκρινίσουμε ότι θα είναι στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο. Κυρία Πρόεδρε, λοιπόν, θα πάψω τώρα και προσβλέπω και στις, στα σχόλια των άλλων ε, συναδέλφων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως σας είπα, έχουμε αρκετούς συναδέλφους που ζητήσαν το λόγο και κάποιοι και νέοι συναδελφοί ήρθαν. Ε, θέλω να ρωτήσω αν οι τελευταίοι αφιχθέντες θέλουν να ε, πάρουν το λόγο. Ο πρώτος, λοιπόν, που θέλει το λόγο είναι ο Πολ Ρανζέλ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες αλλά και τους εισηγητές και να τους συγχαρώ για τη διοργάνωση αυτής της ακρόασης. Και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας των εμπειρογνωμόνων και των συναδέλφων βέβαια σε κάτι που είναι πολύ παράξενο στις δικές σας παρεμβάσεις, ότι δηλαδή συγκρίνετε διαφορετικά συστήματα, αναλύετε τις συνθήκες, αλλά ξεχάσατε την ιστορία. Ποια είναι η ιστορία του Κοινοβουλίου. Είναι μια... Είναι μια ιστορία νόμου νομικήστικη και επιβολής κατά κάποιο τρόπο του Κοινοβουλίου έναντι των καθιερωμένων εξουσιών. Αν δείτε την Αγγλική Επανάσταση 60 χρόνια στον 17ο αιώνα, αν δείτε την Αμερικανική Επανάσταση, αν δείτε την ε, Επανάσταση στη Γαλλική το 1789 βλέπετε ένα κοινοβούλιο που δεν δέχεται τα καθιερωμένα και θεσπίζει τους δικούς του κανόνες για να φτιάξει και να οργανωθεί όπως νομίζει. Ε, εγώ νομίζω λοιπόν πως θα πρέπει να δούμε τα τμήματα, μάλλον τις σχέσεις ε, εξουσιών και μέσα από αυτή την προοπτική μιας, ε, ενός μεταβαλλόμενου συντάγματος και όχι με πολύ νομικίστικο τρόπο. manière juridique. Θα πρέπει να το δούμε, να το εξετάσουμε από συνταγματικό τρόπο. Και θα έλεγα, θα το, το αποκαλούμε δικαίωμα. Ίσως θα ήταν καλύτερα να το πούμε αποκαλέσουμε οργανωσιασιόν σκεφάλ σύμφωνα με τη γερμανική παράδοση οργανωτική εξουσία, ότι δηλαδή το κοινοβούλιο που εκλέγεται θα πρέπει να είναι αυτό που θα έχει και την ε, εξουσία. Γι' αυτό και θα χρησιμοποιήσω τη λέξη ε, του, του δικαιώματος το προνόμιο του διοργάνω, της οργάνωσης. Όχι βασιλικό προνόμιο, αλλά πάντως προνόμιο για οργάνωση. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι όχι μόνο θέμα αποτελεσματικότητας, να βρίσκεται το εκτελεστικό και το κοινοβούλιο στην ίδια πόλη, είναι και θέμα δημοκρατίας. Διότι αν ένα κοινοβούλιο θέλει να ελέγχει το εκτελεστικό της εξουσίας, θα πρέπει να μπορεί και να το κάνει. Αυτή η απόσταση είναι ένας τρόπος αδιαφάνειας. Αυτό που έγινε τα περασμένα χρόνια, ιδιαίτερα μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας, είναι ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει κερδίσει ένα πολύ ισχυρό δημοκρατικό ρόλο. Και επειδή έχει ισχυρό δημοκρατικό ρόλο, πρέπει να έχει και αυτή τη δυνατότητα, την ικανότητα να ελέγξει τις δημοκρατικές δυνάμεις και τις εξουσίες ε, του της Ευρωπαϊκής θα Δεν υπάρχει ίσως η αρμοδιότητα των αρμοδιοτήτων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ως Πορτογάλος θα μπορώ να σας πω ότι πιθανότητα η ιδέα της, κυριαρχία κυριαρχίας να μην είναι τόσο προφανή σήμερα όσο ήταν παλαιότερα. Αλλά όχι μόνο ως Πορτογάλος, πιστεύω ότι από ε, ισχυρές χώρες όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Γαλλία είναι απόλυτα περιορισμένες λόγω του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος. Και για να μιλήσουμε για την αρμοδιότητα των αρμοδιοτήτων ή την κυριαρχία, αυτά είναι λόγια, είναι λέξεις που δεν είναι οι κατάλληλες, δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα των εξουσιών τη σήμερον ημέρα. Αυτό που πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε στο Κοινοβούλιο και αν δεν το, μας το δώσουν θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε και να κάνουμε έκκληση στα ουράνιους υπολόγους στο τελευταίο κεφάλαιο του να βοηθήσουμε το δικαίωμα της μιας έδρας. Δεν μπορεί να είναι το Στρασβούργο, η Βρυξέλλος ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είναι η Βρυξέλλος, όχι επειδή μου αρέσουν ιδιαίτερα, αλλά επειδή εδώ εδρεύουν τα άλλα δύο θεσμικά όργανα, το Συμβούλιο και η Επιτροπή. Και να πω και κάτι ακόμα. Είναι πολύ παράξενο που το Συμβούλιο που είναι ένα είδος δεύτερης βουλής και όχι μόνο αυτό αλλά είναι και ένα όργανο πολι, πολιτικού δικαίου, το πολίτικο όπως λένε οι Ιταλοί, είναι και ταυτόχρονα όμως και μια δεύτερη βουλή. Οι Βρετανοί δέχονται ότι η Βουλή των Λόρδων οι Βρετανοί θα δέχονταν η Βουλή των Λόρδων να αποφασίζει πού θα συνεδριάζει το κοινοβούλιο τους. Το Bundesrag θα πρέπει να αποφασίζει αν το Bundestag θα συνεδριάζει τη Βερολίνο ή όχι. Ε, κάτι τέτοιο θα ήταν απαράδεκτο. Βέβαια, είναι κράτη-μέλη. Δεν έχει νόημα σε ένα από συνταγματική άποψη κάτι τέτοιο. Και αυτό που ήθελα να πω εν τέλει είναι ότι κατά τη γνώμη είναι σαφές πως έχουμε το προνόμιο να ορίζουμε εμείς που θα συνεδριάζουμε. Ακόμα και αν η συνθήκη λέει κάτι άλλο δεν είναι μόνο θέμα των συνθήκων, είναι ένα θέμα των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφόσον εμείς τους αντιπροσωπεύουμε, έχουμε το δικαίωμα να ορίζουμε πού θα συνεδριάζουμε. Ευχαριστώ. The, the, rest of the Ευχαριστώ. προσοχή λίγο στο χρόνο, ε, γιατί θέλει να μιλήσει και ο συνεισηγητής, να απαντήσουν και εμπειρογνώμονες ε, Έχουμε δηλαδή μισή ώρα για όλη αυτή τη συζήτηση, για τους βουλευτές. Και... Ο Γκέραρτ Χέφνερ θέλει να κάνει μια ερώτηση και μετά ο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη. Ε, ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω γερμανικά, μου επιτρέπετε. Για να αξιοποιήσουμε και τους δερμηνείς μας. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ ε, για τις τόσο αξιόλογες παρουσιάσεις σας, ε, θαυμάσιες και πολλοί συνάδελφοι κατάλαβαν ότι λάβαμε υπόψη πάρα πολλά πράγματα κατά την επιλογή των εμπειρογνωμόνων, διαφορετικές σκοπιές, διαφορετικές θέσεις ερευνητών, αλλά και γεωγραφική κατανομή, Γερμανία, Λουξεμβούργο, ε, Βρετανία και Γαλλία. Αυτό που με απασχολεί εμένα και θέλω να ρωτήσω στο τέλος είναι το εξής. Η δημοκρατία στην ιστορία δεν είναι ποτέ κάτι ουρανοκατέβατο ή κάτι που επέρχεται ε, ως φυσικό φαινόμενο. Θα πρέπει πάντα να κατακτάτε ε, και βαθμιαία και σταδιακά. Ποτέ δεν είναι ολοκληρωμένη. Η ιστορία και η εμπειρία μας δείχνει ότι οι κατακτήσεις γίνονται βήμα-βήμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ιστορικό πρότυπο. Από το 1952 δημιουργήθηκε μια κοινοβουλευτική συνέλευση τότε της ΕΚΑΧ για πολύ πρακτικούς λόγους είπαν ότι να συνεδριάζει εκεί που συνεδριάζει το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ε, μετά, από εκεί και πέρα, σιγά σιγά τα διάφορα θεσμικά όργανα ε, προέκυψαν στις Βρυξέλλες και κάποτε φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση. Αυτό το πήγαινε έλα. Βρυξέλλες, Στρασβούργο και οι ρυθμίσει στο άρθρο 341 και ιδιαίτερα το πρωτόκολλο 6 τη συνθήκη. Αν κάνουμε μια ιστορική αναδρομή μπορούμε να τα καταλάβουμε θαυμάσια και να τα εξηγήσουμε. Ε, και πρακτικά όμω, κανεί, αν το δει με ένα Ε, εκπλήσεται γιατί δεν φαϊκό. Και να σας δώσω και ένα παράδειγμα που πηγαίνει πέρα από τη συζήτηση. Πολλοί αναφέρουν συχνά την ε, αποτελεσματικότητα και το έλλειμμα. Δηλαδή εννοούν μόνο το χρόνο και το κόστος που συνδέεται με το ταξίδι αυτό και την απώλεια της ενέργειας και το προσωπικό που ταξιδεύει συνεχώς. Για μένα υπάρχει και ένα άλλο θέμα αποδοτικότητας που το θεωρώ πολύ πιο ε, σοβαρό. Εγώ είχα κάνει τρεις θητείες στη Γερμανική Βουλή πριν έρθω εδώ στο Κοινοβούλιο, όπου θεωρούσαμε πάρα πολύ αυτονόητο να επιμείνουμε το Κοινοβούλιο αν το θεωρεί πολιτικά σκόπιμο να συνεδριάζει σε ολομέλεια μία, δύο, τρεις μέρες μετά από μείζωνα πολιτικά γεγονότα για να έχουμε την ώρα των επίκαιρων ερωτήσεων ή σε μια νομοθετική διαδικασία εντός της εβδομάδας να συγκληθεί το Κοινοβούλιο σε ολομέλεια για να αποφασίσει. Γιατί την ίδια μέρα μπορούμε να έχουμε συνεδριάσεις πολιτικών ομάδων, επιτροπών, διαφόρων ομάδων εργασίας και ολομέλειας. Εδώ επειδή έχω αυτή την πείρα, το βρίσκω πάρα πολύ βαρύ το πλαίσιο, το οποίο απορρέει ε, απλώς και μόνο επειδή κάτι αποφασίστηκε σε μια συνθήκη και μάλιστα όχι από το κοινοβούλιο, δηλαδή τους ανθρώπους που αφορά. Αλλά σε μια συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών που μπορώ να την καταλάβω. Ε, ερωτώ λοιπόν τους εμπειρογνώμονες. Ο ρόλος του κοινοβουλίου με τις διαδοχικές αλλαγές της ε, θήκης, αλλά ιδιαίτερα με τη Λισαβόνα, μήπως έχει αλλάξει όχι μόνο σταδιακά και βαθμία, αλλά και καταρχήν. Και αν είναι καταρχήν αλλαγή ε, του ρόλου του Κοινοβουλίου, αυτό δεν σημαίνει και διαφορετική προσέγγιση στο ζήτημα της έδρας και του χρονοδιαγράμματος, ε, της διάταξης των εργασιών για, απαιτείται κάτι τέτοιο. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλούς τώρα τριμερείς διαλόγους, γιατί είμαστε συνομοθέτες, ε, ισότιμοι με το Συμβούλιο και καλούμεθα να διαπραγματευτούμε. Και με την άδειά σα το βρίσκω λίγο περίεργο να μας ορίζει αυτό το Συμβούλιο με το οποίο είμαστε ισότιμοι που θα συνεδριάζουμε. Είναι περίεργο είναι ε, αυτό μια εξαίρεση για το, του άρθρου 341. Δεν υπάρχει πλέον διαδικασία για το κοινοβούλιο. Ε, είναι τελεσίδικο. Γνωρίζουμε βέβαια τις συνθήκες, αλλά θέλουμε να ρωτήσουμε το Κοινοβούλιο και τους συναδελφούς μήπως χρειάζεται ένα νέο βήμα, όπως έχει διαμορφωθεί πλέον από το νέο ρόλο του Κοινοβουλίου. Δεν είναι πλέον υποχρεωτικό το Κοινοβούλιο να έχει περισσότερη ελευθερία για να ορίζει και το χρονοδιαγραμμά του, άρα και την έδρα του. Εκεί θα μπορούσα να φανταστώ πάρα πολλά πράγματα. Ε, αλλά ε, για μένα το ερώτημα δεν είναι ποιο φαίνεται το τελικό αποτέλεσμα, αλλά είναι συνταγματική η υπόθεση. Γι' αυτό και το συζητούμε εδώ. Επειδή έχει αλλάξει ο ρόλος του Κοινοβουλίου και νομίζω απαραίτητος θα πρέπει να διεκδικήσει αυτό το νέο δικαίωμα το Κοινοβούλιο. Και πώς το φαντάζομαι πολιτικά και νομικά με συντακτική συνέλευση. Και το Κοινοβούλιο να θέσει αυτό το θέμα επιτάπητος, όπως έγινε και στην προηγούμενη συντακτική συνέλευση άλλωστε, και στη διακυβερνητική διάσκεψη. Και θα με παραξέναβε να το απεμβολήσει τώρα το Κοινοβούλιο. Και μια πολύ σύντομη δεύτερη ερώτηση ψάχνουμε προηγούμενα στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι λίγο δύσκολο γιατί έχουμε διαφορετική οργάνωση από ό,τι τα κράτη-μέλη. Και επίσης και για άλλους λόγους δεν υπάρχει ε, προηγούμενο. Το θέμα της πρωτεύουσα σε κάθε κράτος μέλος είναι ιστορικά λιμένο. Ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει τεθεί όμως. Αν τεθεί και ρωτώ τους εμπειρογνώμονες ξανά, ποιος θα κληθεί να αποφασίσει. Παράδειγμα, μιλήσατε για τη Γερμανική Βουλή, Bundestag, αυτό δεν το αποφασίζει μόνο η Κάτω Βουλή, αλλά και η Άνω. Εγώ ήμουν μέλος τη της Κάτω Βουλής όταν αποφασίσαμε για την έδρα μας Βόνη, Βερολίνο και ήταν πολύ μικρή η διαφορά. Και Δης στη Γερμανία, πόσο μάλλον στην ε, κυβέρνηση και ε, σε καμία περίπτωση η Άνω Βουλή δεν ε, θα αμφισβητούσε ότι είναι κυρίαρχο το κοινοβούλιο να το αποφασίσει, χωρίς να το λέει πουθενά το Σύνταγμα. Ποιος άλλος όμως θα το αποφάσιζε αυτό. Ήταν προφανές η ε, συνέλευση, εκλεγμένοι εκπρόσωποι του λαού. Αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν θέλουν να μας παίρνουν σοβαρά υπόψη οι ψηφοφόροι μας. Ευχαριστώ. Τι ερώτηση, βασικά τοποθέτηση ήταν αυτή και ερώτηση. Θα δώσω το λόγο στον Ρομπέρτο Κουαλτιέρη και μετά στο συντονιστή των ε, σοσιαλιστών και μετά στην κυρία Λεγκρίπ. Ε, ε, θα ακολουθήσω και εγώ την συμβουλή του κυρίου Φόξ. Να μην σχολιάσω το έγγραφο εργασία που θα δούμε αύριο, αλλά να προσπαθήσω να υποβάλω κάποια ερώτηση στους εμπειρογνωμονέ μας και να διζητήσω τα δικά του σχόλια για κάποια πράγματα που λέει το έγγραφο εργασίας. Δεν θα ρωτήσω αυτό που με απογοήτευσε ιδιαίτερα, που είναι ένα τεχνικό λάθος στην τελευταία παράγραφο για τη σύγχυση ανάμεσα στην ε, κατακτική απλοποιημένη διαδικασία για την διακυβερνητική συνθήκη. Είναι κάτι και σε σχέση με τα όσα είπε ο Ανδρέας Μάουερ για τα διάφορα είδη διαδικασίες, να πω παρακαλώ μην παρουσιάζετε ένα τέτοιο εγγραφό με πρακτικά και νομικά ασφάλματα. Αλλά για τα πολιτικά θέματα αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω από τους, ε, να, αναπτύξουν οι εισηγητές μας είναι η αξιολόγηση μιας αρχής που κατά τη γνώμη μου λείπει εδώ στο έγγραφο εργασίας και από κάποιες από τις συμβολές της εισηγήσεις. Δηλαδή η αρχική, η ιδιαίτερη φύση της δημοκρατικής νομότητας της Ένωσης με βάση το άρθρο 10 τη διπλή νομιμότητα και τα, τόσο το κράτος μέλος όσο και οι πολίτες αναφέρονται εδώ. Αυτό είναι το αρχικό, αυτό είναι το, αυτή είναι η βάση, η πηγή, η ρίζα και θα μπορούσαμε να ενημερώσουμε, να εξυγχρονίσουμε το πρωτόκολλο 341 γιατί αν λάβουμε υπόψη αυτή την πολύ σημαντική βασική αρχή, αυτό σημαίνει πως ναι, φυσικά το 341 παράγραφος 6 δεν συνάδει με το άρθρο 10 γιατί ζητά και τα δύο και τα κράτη-μέλη και ο λαός να είναι πηγές της δημοκρατικής νομιμότητας αλλά γιατί να πούμε ότι μία, η μία πηγή αποφασίζει για την ίδια μα δεν είναι αυτό το θέμα να λάβουμε υπόψη ότι η βάση είναι ε, ε, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, ο λαός και το Κοινοβούλιο και θα πρέπει να συναποφασίζουν και για το δευτερογενές όσο και για το πρωτογενές δίκαιο. Και δεύτερο θέμα, ερώτημα μάλλον, προς τον κύριο Χόφμαν. Γιατί είπατε 7 από τα 27 συντάγματα. Με εννοείται ότι τα άλλα 21 ότι η απουσία της πρόβλεψης στο Σύνταγμα για την έδρα του Κοινοβουλίου σημαίνει πως το Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει το ίδιο με βάση το δικό του εσωτερικό κανονισμό. Δηλαδή εννοείται ότι το Ιταλικό Κοινοβούλιο αποφασίζει ξαφνικά να μετακομίσει τη Σικελία στο Μιλάνο. Δεν νομίζω πως γίνεται αυτό. Είναι η πρωτεύουσα η έδρα. Εννοείται και αυτό είναι πρωτογενέ ε, δίκαιο, είναι επίπεδο πρωτογενού δίκαιο. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή τι σημαίνει να υποβαθμίζουμε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα στο, στο, επίπεδο του ιστορικού κανονισμού ενό συνταγματικού σώματο. Και εγώ είμαι υπέρ τη μια έδρα, είμαι κατά των δύο εδρών, αλλά πρέπει να αποφασίσουμε ποια θα είναι η στρατηγική. Οπότε και τα δύο στοιχεία είναι πολύ σημαντικά για να διευκρινιστεί το θέμα και αυτό ακριβώς θέλω να ρωτήσω από τους ομιλητές μας. Σας ευχαριστώ και για το ότι τηρήσατε την ώρα και τώρα ο αντιπρόεδρός μας ή αντιπρόεδρός μας. Merci, Madame la, Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να κάνω κάποια σχόλια. Ή ε, να αποπειραθώ να κάνουν και προτάσεις ή ιδέες που να τροφοδοτήσουν ε, επικοδομητικά τη συζήτηση. Πριν από στην ουσία θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο σχόλιο για τη μορφή εντό εισαγωγικών το τύπο μάλλον εντό εισαγωγικών και τη φύση, τη διατύπωση της πρόσκλησης που πέστειλαν οι δυο συνεισηγητές στο σύνολο των μελών ε, του Κοινοβουλίου για να τους καλέσουν να έρθουν να συμμετέχουν στη συναποψινή συνεδρίαση. Νομίζω πω ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε καταρχήν ε, εικονικά όσο και ε, το κείμενο που περιλαμβανόταν σε αυτή την αφίσα για τη σημερινή συνεδρίαση δεν ήταν πολύ ισορροπημένο. Ούτε αμερόληπτο και την, ε, έδινε την αίσθηση ότι χρησιμοποιούσε πολλά από τα επιχειρήματα ή τις οπτικές παρουσιάσεις που έκανε να πιστεύουμε ότι το είχαν σχεδιάσει οι υποστηρικτές της εκστρατείας μια και μόνη έδρα. Η λέξη seat, έδρα, το θέμα του έδρας και του τόπου εργασίας με άφησαν λίγο αμήχανη. Αυτά λοιπόν όπως είπα για τον τύπο. Τώρα, αυτό που είναι σημαντικό επί της ουσίας είναι να δούμε την ευρωπαϊκή ιστορία, να δούμε ότι ε, ε, όσον αφορά την ιστορία της Υπήρους μας και του κόσμου, το ευρωπαϊκό ε, σχέδιο είναι σχετικά πρόσφατο και σύντομο στη διάρκεια του και γεννήθηκε από τη συμφιλίωση ανάμεσα σε λαούς και χώρες που επανελειμμένως είχαν πολεμήσει μέχρι και σε σημείο γενοκτονίας και που κάποια στιγμή αποφάσισαν να φτιάξουν ένα κοινό πρόγραμμα, μια συμμαχία, μια κοινότητα ζωής και μέλλοντος, ένωση οικονομική και πολιτική που ήταν τελείως πρωτότυπη, είναι τελείως ένα οικοδόμημα sui generis ιδιόμορφο και ανταποκρίνεται στην απόπειρα οικοδόμησης κάποιου κάτι νέο που δεν έμοιαζε με τίποτα που υπήρχε στα εγχειρίδια συνταγματικού δικαίου ή αλλού στον κόσμο. Δεν είναι ομοσπονδία, δεν είναι συνομοσπονδία, δεν είναι ούτε και το συνέδριο της, της Βιέννης που θέλουμε εδώ τώρα να ξαναζήσουμε, αλλά είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και το, τα ίδια χαρακτηριστικά λοιπόν, αλλά και η πρόσφατη ιστορία, ε, μας οδηγούν στο να σκεφτούμε ότι οι νομικές και συνταγματικές ιδέες που μπορεί να κυριαρχούν σε άλλες ανθρώπινες μορφές ή θεσμούς δεν μπορούν να άμεσα να μεταγραφούν. Και εφόσον πρόκειται για ένα πολιτικό οικοδόμημα που δεν είναι σε αυτό το στάδιο, ορισμένοι βέβαια πολλοί θα το ήθελαν, αλλά πάντως διαπιστώνουμε σε αυτό το στάδιο δεν είναι ένα ομοσπονδιακό κράτος αυτό το πολιτικό οικοδόμημα, οτιδήποτε μπορεί να μοιάζει με συγκέντρωση των χώρων, των τόπων εξουσίας δεν θα πρέπει να γίνει, ε, κατά τη γνώμη μου και για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι συζητήσεις εδώ και πολλά χρόνια εδώ στο Κοινοβούλιο και πιο πρόσφατα και στο, εδώ στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων φαίνεται να υπάρχει βούληση να προχωρήσουμε προς μια ομοδοποίηση, προς μια μάλλον συγκέντρωση σε ένα συγκεκριμένο τόπο εργασίας για τις δραστηριότητες του Ευρωκοινοβουλίου, δηλαδή ένα είδος και συγκέντρωσης και της δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής πρωτεύουσας ε, κατά τη γνώμη μου ωστόσο αυτό δεν αντιστοιχεί στην φύση αυτού του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, του αρχικού, που όπως είπαμε είναι sui generis. Ευρωπαϊκό οικοδόμα είναι ένα οικοδόμα δικαίου. Έχουμε δηλαδή μια κατάσταση συγκεκριμένη, ξεκάθαρα κείμενα, τις συνθήκες, τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που με μεγάλη σαφήνεια έχω την εντύπωση θυμίζουν τη διασύνδεση ανάμεσα στις αρμοδιότητες των κρατών μελών και του Κοινοβουλίου όσον αφορά την εσωτερική διοργάνωση των εργασιών του και υπάρχει μια λεπτή ισορροπία η οποία έχει εξευρεθεί και εκεί η αποφάση του ΔΕΚ την πλαισιώνουν αυτή την διπλή πολιτική νομιμότητα της οικοδόμησης της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. εκπροσωπούνται οι πολίτες αλλά και τα κρατημέλη Και νομίζω πως είναι σημαντικό να συνεχίζουμε να αναζητούμε με ποιο τρόπο θα σεβαστούμε αυτή τη λεπτή ισορροπία. Αυτά. Δεν θα πω τίποτα άλλο, αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι κάθε πολιτικό οικοδόμα εντάσσεται σε ένα ιστορικό πλαίσιο που αποτελεί και τον πλούτο και την ιδιαιτερότητά του. Of course, as uh, we are the only speaker as a woman, that's why you... Βέβαια μόνη γυναίκα, γι' αυτό σας αφήσαμε, μιλήσετε λίγο παραπάνω, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δεν μπορεί όλος ο, ο κόσμος να μιλάει το ίδιο. Λοιπόν, παρακαλώ τον Αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου να πάρει το λόγο, τον κ. Μακμήλαν Σκότ και μετά ο κ. Ρούτσας. Ε, Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε. Πραγματικά ενδιαφέρουσα συνάντηση και συγχαρητήρια στους εμπειρογνώμονες. Ως Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου έχω να πω ότι το Προεδρείο που είναι αρμόδιο για οικονομικά και οργανωτικά θέματα, ούτε το ίδιο το Προεδρείο μου, ούτε το ίδιο το Κοινοβούλιο έχουν διεξαγάγει συζήτηση για τους τόπους εργασίας για πολλά χρόνια. Θεωρώντας λοιπόν ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο να γίνει, έφτιαξα το 2010 μια μικρή ομάδα, θεωρώντας ότι οι ευθύνες που αναλαμβάνει το Κοινοβούλιο γίνεται όλο και πιο δύσκολο να τις αντιμετωπίσουμε έχοντας να δουλέψουμε σε δύο ή και τρεις έδρες εργασίας. Αυτή λοιπόν η μικρή ομάδα ανέλαβε την εκστρατεία της μιας έδρας. Έχουμε μια μικρή steering group 20 περίπου ευρωβουλευτών από διάφορες πολιτικές ομάδες. Παρακολουθούμε τις ψηφοφορίες και τις καταγράφουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι εμπειρογνώμονες σας μίλησαν για δημοσκοπήσεις που έκανε η European Research Group, γιατί παρακολουθούν και καταγράφουν τις γνώμες των βουλευτών. Όμως οι πιο συγκεκριμένες αλλαγές εμφανίζονται από τις ψηφοφορίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο και σας παραπέμπω στην ιστοσελίδα μας singleseat.eu το 2013 78% για την ψηφοφορία του προϋπολογισμού 78% των ευρωβουλευτών ζήτησαν από τις κυβερνήσεις να επανεξετάσουν το θέμα των εδρών 74% ζήτησε έναν οδικό χάρτη με χρονοδιάγραμμα προς την κατεύθυνση μιας μονής, μιας μοναδικής έδρας. Υπάρχει λοιπόν μια σημαντική πλειοψηφία που ζητεί αλλαγή. Και αυτό είναι σημαντικό. Το είπαν και οι δύο εισηγητέ, αλλά και η Επιτροπή Αναφορών που συνέρχεται αύριο για παρόμοιο θέμα και κοιτάζει το 1,7 εκατομμύρια πολίτες που απευθύνουν αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο πρόεδρος Σούλτ τη δέχθηκε ως παραδεκτή. Πολύ, αυτά λοιπόν πολύ σύντομα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναφέρθηκε στην ε, περίοδο συνόδου ψηφοφορίας του προπολογισμού του Κοινοβουλίου σαν να έχει κάποιο ειδικό καθεστώς. Αυτό δεν συνισχύει πλέον όμως. Είδαμε άλλωστε τους τελευταίους μήνες βαθιές αλλαγές από το ίδιο το Συμβούλιο. Υπάρχει διάταξη τη συνθήκης που λέει ότι τρεις φορές το χρόνο το Συμβούλιο συνέρχεται στο Λουξεμβούργο. Τον Απρίλη έγιναν πολλές συνεδριάσεις στο Δουβλίνο του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο λοιπόν συναπαρτίζεται και σε ορισμένε μορφέ το από πολλά χαρτοφυλάκια. Αλλάζει λοιπόν τον τρόπο εργασία του. Το Ευρωπαϊκό Δε Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά εδώ στι Βρυξέλλε όταν το Κοινοβούλιο συνέρχεται σε περίοδο συνόδου στο ε, Στρασβούργο. Σε αυτή λοιπόν την δίθεν δημοκρατική διαδικασία φαίνεται καθαρά πόσο χαμηλή άποψη έχει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. η πλειοψηφία αυτή των Ευρωβουλευτών που ανέφερα πριν δεν έχει καμία, κανένα συνταγματικό καθεστώ. Όμω πρόκειται για μια σημαντική πλειοψηφία, 74 ή 78% των βουλευτών. Δεν μπορεί να αγνοηθεί. Εν τέλει, το θέμα θα, στο θέμα θα δοθεί πολιτική και όχι διπλωματική λύση. Τώρα το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ζητήσει να αναλάβει την έξτρα ευθύνη, την ικανότητα για να αποφασίσει πού και πότε θα συνέρχεται. Ευχαριστώ και ευχαριστώ που τηρήσατε το όριο χρόνο σας. Ο κύριος Δρούτσας, άλλος κανείς αν επιθυμεί να λάβει το λόγο. Εσείς, κύριε Νταφ, οκ. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομος διότι τα περισσότερα από τα θέματα ήδη τέθηκαν και από τον μόλις προλαλήσαντα. Η ερώτησή μου, ωστόσο, ευθυγραμμίζεται και με εκείνη του κυρίου Χέφνερ σχετικά με τις επιπτώσεις στη νομική κατάσταση με την αλλαγή του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου που γίνεται ένας πραγματικός συνομοθέτης. Και δεύτερο, αυτά που εξήγησε ο καθηγητής Κώστα και που άλλωστε τα επανέλαβε ο προηγούμενος ομιλητής, εσείς συνοψίσατε όλη την υπόθεση σε μια φράση. Όλες οι συζητήσεις που διεξάγουμε εδώ, εντός του σώματος ή αλλού, όλες κατευθύνονται στην κατεύθυνση αυτή και μπορούν να συνοψιστούν ως εξής το θέμα τη έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορεί να ρυθμιστεί παρά μόνο πολιτικός. Είναι πολιτικό θέμα. Είναι πολιτικό θέμα. είμαστε ειλικρινεί και είμαστε σαφεί. Γι' αυτό και θα ήθελα να σα ρωτήσω ένα άλλο πράγμα ε, σχετικά με μια άλλη προσέγγιση. Επειδή έχουμε τι εμπειρίε του παρελθόντο με χώρε μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβούλιο που αγνοούν το θέμα αυτό. Ακόμα και η αναφορά που αναφέρθηκε πριν και που έχει υπογραφεί με, από πάνω από 1,2 εκατομμύρια πολίτες αγνοείται τι μπορεί να γίνει λοιπόν παραπάνω έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δεχτεί να το εγγράψει στην ατζέντα του. Δηλαδή τι μπορεί να κάνει η ίδια η κοινωνία, ο ίδιος ο Ευρωπαίος πολίτης. Ας πούμε σε ένα πανευρωπαϊκό δημοψήφισμα μπορεί κάτι τέτοιο να αποτελέσει λύση, μια λύση που θα μπορούσε να μας βοηθήσει, να μας στηρίξει σε αυτή την κατεύθυνση. Ας είμαστε ρεαλιστές. Θα υπάρξει τουλάχιστον πάντα ένα βέτο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το θέμα αυτό, έτσι δεν είναι. Και μια και έχω ακόμα ένα-δύο λεπτά, ήθελα να πω ένα πράγμα ακόμη. Αυτή η δίθεν ιστορικο-συμβολική αξία του Στρασβούργου. Βεβαίω είναι η αληθέ και είναι σημαντική. Α μην, μην τη λησμονούμε, αλλά α μην λησμονούμε ακόμη και την σημερινή πραγματικότητα. Η σημερινή πραγματικότητα είναι μια βαθιά οικονομική κρίση και ένας αυξανόμενος ευρωσκεπτικισμός. Θέματα όπως η έδρα του Ευρωκοινοβουλίου μέσα στην τρέχουσα αυτή κατάσταση, δυστυχώς, ας είμαστε λοιπόν και εδώ σαφείς και ειλικρινείς, ένα από τα κύρια επιχείρηματα, ένα εύκολο λαϊκίστικο επιχείρημα, το οποίο στρέφεται κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπα, σε τόσο δύσκολη περίοδο για την Ένωση. Ασφαλώς λοιπόν η ιστορική συμβολική αξία του Στρασβούργου πρέπει να διατηρηθεί, αλλά ίσως θα πρέπει να αναρωτηθούμε ή να σκεφτούμε περισσότερο, να προβληματιστούμε περισσότερο, με ποιον άλλο ίσως τρόπο μπορούμε να τονίσουμε αυτή την συμβολική αξία. Δεν είναι απαραίτητο να είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκεί. Μπορεί το Στρασβούργο να γίνει η έδρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο κύριος Μάουρερ είπε ε, ε, ε, για μια στιγμή έδειξε για μια διαφάνεια, ίσως να είναι χρήσιμο και εμάς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προβληματιστούμε περισσότερο επί μια εναλλακτική προτάσεως για το Στρασβούργο. Έτσι ώστε να έχουμε στη διάθεσή μας πλέον πιστικά επιχειρήματα που να μπορέσουμε να την παραβάλουμε απέναντι σε ορισμένες χώρες μέλη. Εσείς τώρα ο κύριος Μπρόνς. Θα κάνω κάτι που συνήθως δεν πρέπει να κάνει κανείς στην πολιτική. Ε, να κάνεις μια ερώτηση που όχι μόνο δεν ξέρεις την απάντηση, αλλά που θα έπρεπε να την ξέρεις. Όταν οι Βρυξέλλες προσωρινά το 2008 εχθρίστηκαν ενιαία έδρα, ποιο ήταν τότε το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε. Δηλαδή προβλέπετε κάποια επίγουσα ανάγκη στις συνθήκες. Αν μπορώ να συνοψίσω εγώ, όχι σωστά βέβαια, τους ε, ε ομιλητές, μας έδωσαν πολλά ε, ε, παραδείγματα για τον τρόπο που δεν ορίζουν τα κοινοβούλια την έδρα τους. Και ιστορικά δεν γίνεται αυτό, εκτός αν έχουμε οι μη επαναστατικές καταστάσεις. Εγώ δεν είμαι υπερενθουσιώδης ούτε για το Κοινοβούλιο γιατί για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτιμώ ένα Κοινοβούλιο χαμηλού κόστους περισσότερο από ότι υψηλού κόστους. Και παρότι το Στρασβούργο που σε πολλές, από πολλές πλευρές ε, είναι προτιμότερο από τις Βρυξέλλες ε, η εύκολη λύση θα ήταν οι Βρυξέλλες γιατί είναι πιο εύκολο να φτάσει κανείς εδώ. Αυτό που είπε ο κύριος Ράγγελ για το ρόλο του Κοινοβουλίου να ελέγχει την εκτελεστική εξουσία είναι πολύ πιο εύκολο όταν είσαι σε διπλανά κτίρια ή στο ίδιο κτίριο ακόμα και για την συνομοθετική μας ε, δραστηριότητα και τέλος και είναι καλύτερη και η στέγαση των βουλευτών στη Βρυξέλλες. Στο Στρασβούργο είναι τα θέματα πάρα πολύ πιεσμένα. Και γενικότερα η νομοθεσία είναι ένα συλλογικό έργο. Ευχαριστώ πολύ. Και ο κύριος Νταφ τελευταίος. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ε, υποτιμώ ούτε παραβλέπω καθόλου το ιστορικό στοιχείο που συζητήσαμε και θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε περισσότερο, αλλά αν στραφούμε προς το μέλλον, γνωρίζουμε όλοι ότι το θέμα αυτό της έδρας δεν μπορούμε να το δούμε ξεκομμένο από πάρα πολλά άλλα θέματα και απομονωμένο. Και το 2015 ε, την Άνοιξη. Νομίζω και είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα γίνει μια ε, συντακτική συνέλευση με ευρύτατα ε, θέματα και πολύ μεγάλη ημερήσια διάταξη από συνταγματικής πλευράς και μεταξύ άλλων θα ορίσει και ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Δημοσιονομικής Ένωσης. Και είτε αρέσει αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε δεν της αρέσει, που μάλλον δεν θα της αρέσει, ε, θα είναι ε, ένα σώμα που θα μετατραπεί σε μια διακριτή και λειτουργούσα κυβέρνηση. Δηλαδή, ο πολιτικός έλεγχος του Κοινοβουλίου ε, θα είναι πιο στενός και πιο κοντινός προς την εκτελεστική εξουσία από ό,τι σήμερα. Ένα δεύτερο που θα κληθεί να κάνει είναι αυτή η, ε, η συντακτική συνέλευση, είναι λογικά να επιφέρει μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ ε, των διαφόρων ε, νομοθετικών σωμάτων. Δηλαδή, Ποια είναι η λογική. Δεν πρόκειται το κοινοβούλιο να είναι σε θέση να αποφασίσει για την έδρα του, αλλά θα πρέπει με κάποιο τρόπο, αν ε, γίνει μια αλλαγή, να επιτύχει τη συμφωνία του Συμβουλίου. Δηλαδή, πολύ μεγαλύτερη εστίαση από ό,τι ποτέ στο παρελθόν θα τεθεί στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας. Δηλαδή, την αρχή που λέγει ότι τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να σέβονται το ένα το άλλο και να συνδράμουν το ένα το άλλο στην εκπλήρωση των στόχων της συνθήκης. Και θα παρακαλούσα τους εμπειρογνώμονές μας να σκεφτούν με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε μια ε, πιο έντονη έκφραση αυτής της αρχής της ειλικρινούς συνεργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω την ευκαιρία σε όλους τους εμπειρογνώμονες να απαντήσουν. Πέντε λεπτά έκαστος και να αρχίσουμε την αντίστροφη σειρά. Πρώτος ο κύριος Μάουρε, γιατί νομίζω έτσι ήθιστε. Ναι. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και τις ερωτήσεις. Ε, θα τις απαντήσω όλες, δεν θα απαντήσω επιλεκτικά. Πρώτον, ε, να αρχίσω από το τελευταίο σχόλιο του Άντρου Νταφ. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ε, να δούμε τι θα ζητήσει το Κοινοβούλιο. Θα πιέσει για αλλαγή της οργάνωσης, της έδρα. Αν το κάνει αυτό, δεν θα γίνει ξεκομμένο θα είναι ένα ε, στοιχείο μόνο μιας ευρύτερης συντακτικής συνέλευσης. Και για να συγκρουστεί με το Συμβούλιο νομίζω δεν αρκεί το θέμα της έδρας. Υπάρχουν πολλά άλλα θέματα. Ε, θα επανέλθω σε αυτό και ε, σε ένα σχόλιο προς τον κύριο Γκολτιέρη. Σε μια μελλοντική συντακτική συνέλευση το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να πείτε εξή το άρθρο 41 ε, και το άρθρο 10 δεν αντιστοιχούν, δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Γιατί? στην περασμένη Ευρωπαϊκή Συντακτική Συνέλευση δεν το έκανε ζήτημα αυτό η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου. Δεν επικεντρώθηκε σε αυτό γιατί ήταν πολλά τα άλλα ζητήματα. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να θέτει και προτεραιότητες και να επιλέγει το Κοινοβούλιο. Και προτεραιότητες σημαίνει ότι αναγνωρίζεις ότι κάποιο θέμα είναι σημαντικό και κάποιο άλλο είναι ίσονος σημασίας. Αν αυτό το θέμα είναι η μέγιστη μεταρρύθμιση. Υπάρχει ε, ο εκδημοκρατισμός της ΩΝΕ, της ΚΕΠΑ, της ΕΠΑ και άλλων θεμάτων. Αν η, βασική προτεραιότητα αυτή, καλώς, αλλά να το αποφασίσετε. Και επίσης το θέμα της διπλής νομιμότητας πολιτών και κρατών θα πρέπει κάπως να μεταφραστεί σε μία απόφαση. Ίσως να πούμε ότι προχωρούμε στη μεταρρύθμιση του άρθρου 48, εδάφιο 3, ε, δεύτερη φράση της ε, ε, τακτικής απλουστευμένης διαδικασίας για τη συναπόφαση στο πρωτογενές δίκαιο. Αν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ότι υπάρχει ένα μικρό τμήμα του πρωτογενούς δικαίου, ένα κλάσμα, ξέρω εγώ, διοργανικό πρωτογενές δίκαιο για τα οργανωτικά θέματα, που είναι αντικείμενο συναπόφασης ε, μεταξύ Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με κόκκινε γραμμέ από εθνικά κοινοβούλια και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια επιλογή για να το συζητήσει καν το Λουξεμβούργο και η Γαλλία. Αλλιώ δεν έχει ε, κανένα μέλλον. Ε, απαντώ στα γερμανικά στα σχόλια του κυρίου Χέφνερ. Εγώ δεν θα χρησιμοποιούσα ως επιχείρημα τους τριμερείς διαλόγους ε, από τη Λισαβόνα. Γιατί οι τριμερείς διάλογοι μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη αποδοτικότητα, αλλά πολύ μικρή διαφάνεια. Και δεν είναι επιχείρημα αυτό για να φύγει από το Στρασβούργο το κοινοβούλιο. Εγώ θα το κρατούσα αυτό απ' έξω. Είναι πάρα πολύ αποτελεσματική ε, η τριμερείς διάλογοι αλλά δεν ε, είναι επιχείρημα για το κοινοβούλιο ούτε από τη βιβλιογραφία αυτό. Είναι ένα επιχείρημα των μεγάλων, των ισχυρών, των πλουσίων και του Συμβουλίου. Το κοινοβούλιο χρειάζεται αυτονομία και μπορεί ε, να χρειάζεται να αποσύρεται κάποιο διάστημα να το συζητάει μεταξύ του. Και κύριε Ρανζέλ, εγώ δεν θα μιλούσα για το Μυραμπό ούτε για την Γαλλική Επανάσταση. Έχουμε μια διαδικασία που είναι μια συνεχιζόμενη αλλαγή και μεταρρύθμιση. Είναι πολύ πιο δυναμική η διαδικασία από ό,τι στα κράτη-μέλη. Η προσαρμογή δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα νέα δεδομένα. Αυτό που χρειάζεται είναι μια δέσμη μέτρο, ένα πακέτο για τη μεταρρύθμιση που να μπορούν να αποφασίζουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Το θέμα δεν είναι μόνο το Συμβούλιο ή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απέναντι στο Κοινοβούλιο. Το άρθρο 341 ορίζει πάρα πολύ ξεκάθαρο ρόλο για τα κράτη-μέλη. Δηλαδή δημιουργεί ε, μια ιδιότυπη διακυβερνητική διάσκεψη που δεν υπάρχει ουσιαστικά, εδώ όμως υπάρχει. Ας πούμε, στην εκπαιδευτική πολιτική τη δεκαετία του 80 είχαμε κάτι τέτοιο. Διαρκής ε, διακοινοβουλευτική διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού ή Παιδείας. Αυτό έχει καταργηθεί. Εδώ παραμένει. Ε, αν μη τι άλλο χρειάζεται τροποποίηση και να μην είναι τα κράτη-μέλη, αλλά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή διάφοροι σχηματισμοί του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χόφμαν. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να πω φυσικά ότι ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη την ιστορική πλευρά, το χειραφέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την αύξηση, τη μεγάλη αύξηση εξουσιών ε, διαχρονικά απέναντι στα άλλα θεσμικά ε, όργανα, αλλά και ταυτόχρονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και μάλιστα, όπως είπε και ο κ. Χόφμα, σε πολλούς τομείς όπου το Κοινοβούλιο πρέπει να ε, πάρει περισσότερες εξουσίες, που είναι πολύ σημαντικό για την νομιμότητα της διαδικασίας στην Ένωση. Αλλά και πρέπει να δούμε και ποια είναι τα γεγονότα, τι ισχύει. Δηλαδή, είναι μια ένωση υπό το κράτος δικαίου και έχουμε κάποια συγκεκριμένη συνταγματική δομή σύμφωνα με τις συνθήκες που όχι μόνο ορίζει ποιος έχει το δικαίωμα να αποφασίζει αυτά τα θέματα αλλά επίσης περιγράφει ακριβώς πώς γίνεται και εκεί ακόμα και στη διαδικασία τροποποίησης των συνθήκων στο τέλος είναι η διακυβερνητική που ορίζει με κοινή συμφωνία ποιες αλλαγές θα γίνουν στις συνθήκες ακόμα και αφού θα έχει εκφέρει τη γνώμη της η συνέλευση. Αυτό ισχύει και δεν μπορούμε να παρακάμψουμε τόσο εύκολα τα κρατημέλη. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να γίνει, κατά τη γνώμη μου για το Κοινοβούλιο, είναι να έχει μια στρατηγική τόσο βραχυπρόθεσμη και ίσως και όσο, όχι και τόσο βράχη η ή μακροπρόθεσμη και μια μακροπρόθεσμη ιεράρχηση προσεγγίσεων που μπορεί να είναι είτε να διαγραφούν οι κανόνες αυτοί τελείως, το πρωτόκολλο 6 και το 341 που αφορά το Κοινοβούλιο, πράγμα που με τη σειρά του θα σήμαινε ότι ε, τα δικαιώματα του κοινοβουλίου, θα είναι αυθύπαρκτα και μεταξύ αυτών και το δικαίωμα στην διοργάνωσή του, στην οργάνωση λειτουργίας του και έπειτα ή διαφορετικά να έχουμε μια ανάλυση, μια ολόκληρη σειρά άρθρων που θα αφορούν ε, την ειλικρινή συνεργασία, που θα αφορούν ε, την ιδέα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και μέσω της αντιμετώπισης αυτού του πακέτου άρθρων της Εθήκης να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα για το Κοινοβούλιο και την ενίσχυση της δημοκρατίας. Αλλά σε όλα αυτά βεβαίως Εάν κανείς ρεαλιστικά δει το θέμα, και αυτό αναφέρθηκε επίσης, θα πρέπει να λάβει υπόψη κανείς την ιστορική εξέλιξη του Κοινοβουλίου και της ε, Ένωσης εν γέννη, για να δει τι μπορεί να γίνει και τι πρέπει να γίνει για να αντικατοπτρίζεται η διαφορετικότητα και η διόμορφη φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι ένα κράτος μέλος. Και για την τελευταία σας ερώτηση να πω ότι στα συντάγματα των 100 μελών υπάρχουν πραγματικά ενδιαφέροντα ενδιαφέρουσες διαφορές σε κανόνες. Στα 16 κράτη-μέλη έχουμε τις διατάξεις για την πρωτεύουσα, 6 συντάγματα που αφορούν την έδρα του Κοινοβουλίου. Στα 17 ε, ε, υπάρχουν συνταγματικές διατάξεις για τις ε, κοινοβουλευτικές συνόδους. Στα 24 κράτη, μάλλον συντάγματα των κατώμενων υπάρχουν διατάξεις που ρητά δίνουν στο Κοινοβούλιο το δικαίωμα να θεσπίσουν τον ιστορικό τους κανονισμό. Ε, υπάρχουν λοιπόν μεγάλες αποκλήσεις αλλά υπάρχει και ένα δεδομένο πλαίσιο για το δικαίωμα στην οργάνωση. Δεν νομίζω δε πως με το παράδειγμα μιας επανάστασης θα μπορούσαμε με τον καλύτερο τρόπο να λύσουμε το θέμα καλύτερα, να δούμε ποιος αποφασίζει γιατί και τι ισχύει πραγματικά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ εσείς τώρα. Ναι, δεν θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά σε ορισμένες. τι να κάνουμε με τα άρθρα της συνθήκης. Αν μπορεί να γίνει με απλό τρόπο. Αυτό πρέπει βέβαια να ενταχθεί μέσα σε ένα πλαίσιο θεμάτων. Νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε είναι ιστορικός. Και παλαιές εξαρτήσεις που ενδεχομένως περιορίζουν το τι μπορεί να κάνει κανείς αργότερα. Ίσως βρισκόμαστε τώρα σε διαφορετική κατάσταση και ο κύριος Χέφνερ, είναι σωστό αυτό που λέει, το κοινοβούλιο έχει μεταμορφωθεί από αυτό που ήταν όταν άρχισε η, ε, η, πορεία της κοινότητας τότε με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακος και Χάλιβος. Αυτό που είδαμε είναι μεγάλες αλλαγές στην νομοθετική ουσία του Κοινοβουλίου και βεβαίως αλλαγή στις διαδικασίες του. Ορισμένες όμως δεν προχώρησαν πολύ, κυρίως για την έδρα εργασίας του, τον τόπο εργασίας του αυτή η διπλή νομιμοποίηση είναι σημαντική. Αλλά είναι κάπως ασυνήθιστο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Διότι οι χώρες μέλη δεν αποφασίζουν επί του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο τρόπος, ωστόσο, του εργασίας του Κοινοβουλίου και ο τόπος είναι τόσο στενά συνδεδεμένος με τον τρόπο εργασία του και τον κανονισμό του επομένω, που δεν είναι παράξενο να επιτρέψουν οι χώρε μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφασίζει το ίδιο. Και δεν είναι ασύνηθε αυτό για ένα κοινοβούλιο το οποίο δεν είναι ακριβώ βέβαια μέσα σε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνηση. Η διαμόρφωση, η τρέχουσα διαμόρφωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπαίνει σε κανένα μοντέλο, αλλά σαφώ δεν είναι κοινοβουλευτικό σύστημα. Η Κομισιόν είναι εκτελεστική εξουσία δεν έχει τη δυνατότητα να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνη, για παράδειγμα, για να αναγκάσει του βουλευτέ να ψηφίσουν με τον αρθίτο τρόπο, αντίθετα από κυβερνήσει που λειτουργούν μέσα σε κοινοβουλευτικά συστήματα. Επομένω, το Κοινοβούλιο έχει βεβαίω μεγάλη ελευθερία και το να αποφασίσει το πού τοποθετεί την έδρα των εργασιών του είναι τόσο στενά συνδεδεμένο με τον τρόπο λειτουργία του που θα έπρεπε να του επιτραπεί. Όπω είπα βέβαια και πριν, το ζήτημα είναι πολιτικό και άρα δεν υπάρχει εύκολη λύση διότι δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να το αποφασίσει ή να το υλοποιήσει με μια απλή αναθεώρηση της συνθήκης. Α, ναι, ναι. Υπάρχει και μια άλλη ερώτηση του κύριου Δρούτσα για το πώς μπορούμε να βάλουμε το θέμα, να αγκάσουμε το, δηλαδή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγγράψει το θέμα στην ατζέντα του. Κάτι που έδειξαν οι έρευνες για τις ευρωεκλογέ είναι ότι αυτές στρέφονται συχνά γύρω από εθνικά θέματα και όχι τόσο γύρω από ευρωπαϊκά. Υπάρχει και ένας μικρός αριθμός ενδείξεων ότι και ε, τα ευρωπαϊκά θέματα έχουν κάποια επιρροή στην έκβαση των ευρωεκλογών και κυρίως των τελευταίων. Αυτό ωστόσο ίσως αποδειχθεί ένα θέμα που θα παίξει ένα ρόλο ίσως στις επόμενες ευρωεκλογές με υπερεθνικές ομάδες κομμάτων που θα υποβάλουν υποψηφιότητες για την Προεδρία της Κομισιόν και ίσως με αυτόν τον τρόπο να υπησέλθει και το θέμα του τρόπου οργάνωση των εργασιών του Κοινοβουλίου στην προεκλογική εκστρατεία. Γκουρμάι. Α, θέλετε ένα σχόλιο. Α, μια ερώτηση κύριε Γκουαλτιέρη. Ναι, μα κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Να γίνει μια διάκριση δηλαδή, αν υπάρχει, ανάμεσα στην αυτοδιάθεση ε, του κανονισμού και της έρας. 27 χώρες μέλη. Ανάμεσα σε αυτές. Σε πόσες από αυτές το Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει το Κοινοβούλιο το ίδιο που θα τοποθετήσει την έδρα των εργασιών του. Με δική του απόφαση. Και το άλλο με, η άλλη επιλογή θα ήταν δηλαδή με νόμο. Αυτό είναι σημαντικό για μας για να έχουμε την εικόνα των διαφόρων επιλογών που υπάρχουν ας πούμε στο συνταγματικό επίπεδο. Μάλιστα, σας ευχαριστώ λέει η Ζήτα Γκουρμάη. Ναι, ωραία θα είναι αν μπορείτε να αποφασίσετε. Να, συγγνώμη, να απαντήσετε. Ο κανονισμός ε, λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν θέλετε, ιεραρχικά ε, τοποθετείται περίπου στο ίδιο επίπεδο με τις νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νομίζω όμως ότι υπό την έννοια αυτή ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήταν σημαντικό να γίνει μια διαφοροποίηση. Και στα κράτη-μέλη είναι πολύ διαφορετικά τα μοντέλα που ισχύουν. Εγώ σας έδωσα έτσι μια πολύ αδρή εικόνα με, με τα αριθμητικά στοιχεία ότι υπάρχουν συντάγματα που το προβλέπουν. Βέβαια, αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι απουσία ρητής ε, αναφοράς στο Σύνταγμα, η αρχή της αυτοργάνωσης θα έδινε την εξουσία αυτή σε ένα κοινοβούλιο. Αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο. Ενδεχομένω θα μπορούσε κάποιο να φανταστεί ότι η απουσία κανόνων θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω αν θα ήταν αυτό το πιο εύκολο να επιτευχθεί, αλλά... Λέτε ότι το 72% επιλέγουν ε, τις Βρυξέλλες. Αυτά τα στοιχεία τα γνωρίζουν και στις διάφορες πρωτεύουσες των κρατών μελών. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα τελευταίος ο κύριος Κώστα. Ευχαριστώ για την προσέγγιση μας. Νομίζω ο καθένας έχει την ε, δική του προσέγγιση. Είμαστε εδώ σε Προσπαθούμε να είμαστε ρεαλιστές και να εξετάσουμε το θέμα και να το σκεφτούμε στα πλαίσια των συνθήκων και των συνταγμάτων. Δεν ξέρω αν θα κάνει επανάσταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό ελέγχεται. Ε, δεν θέλω να το συζητήσω. Πάντως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει καμιά ιδιάζουσα θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που συνδέεται με αυτή τη δυναμική. Ορισμένοι όπως ο Ρίτσαρτ Κόρμπετ περιγράφουν ότι αποκτά όλο και περισσότερες εξουσίες και μπορεί κάποια στιγμή να διεκδικήσει το δικαίωμά του να διοργανώνει ή να οργανώνει τις εργασίες του. Αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα όμως. Χρειάζεται να θεώρηση τη συνθήκη ε, που κατά κάποιο τρόπο επιβάλλεται. Αν γινόταν κάτι τέτοιο, το κοινοβούλιο αυτό θα ήταν ισχυρότερο από οποιοδήποτε άλλο εθνικό κοινοβούλιο. Θα ήταν υπερομοσπονδιακό κοινοβούλιο πάρα πολύ ισχυρό που δεσμεύεται από πολλή στοιχεία στη συνθήκη ε, ε, αλλά χωρίς δημοκρατική τέτοια νομιμότητα, γιατί κανείς δεν μπορεί να το διαλύσει το κοινοβούλιο και να ζητήσει προώρες ευρωεκλογέ. Και ποιο κράτος θα δεχόταν τέτοιες υπερεξουσίες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για το θέμα της κινητοποίηση των πολιτών που έθεσε ο κύριος Ρούτσας, ε, να προκαλέσω λίγο, αν συμφωνείτε έτσι να σας προβοκάρω λίγο, νομίζω δεν θα πρέπει να υπερεξουσίες υπερτιμούμε την ε, κινητοποίηση των πολιτών. Εντάξει, η αναφορά με 1,2 εκατομμύρια υπογραφές αυτό είναι τεράστιο επίτευγμα. Αλλά εγώ εργάζομαι ε, πάνω από 20 χρόνια επί των θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχω εργαστεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ξέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα της έδρας για οποιονδήποτε εργάζεται εδώ, για τη ζωή του, για τη διαβίωση του. Οι υπόλοιποι πολίτες εκτός ε, δεν ανησυχούν και τόσο πολύ όσοι γνωρίζουν καν αυτό το θέμα έτσι. Και αν έχει αρνητική επίπτωση το επιχείρημα αυτό της έδρα στους πολίτες, αυτό το χρησιμοποιούν οι ευρωβουλευτές, ούτε οι πολίτες ούτε το μέσο, το μέσο ενημέρωσης. Υπάρχουν άλλα που μπορούν να σκανδαλίσουν τους πολίτες για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την ευρωπαϊκή πολιτική εν γέννη. Συμφωνώ πολύ με τους συναδέλφους λοιπόν που λέγουν ότι ρεαλιστική λύση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήταν να ζητήσει νέα διαπραγμάτευση για τη συνθήκη συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων της Έδρα μέσα σε ένα συνολικό πακέτο, έτσι μια δέσμη ε, προσυμφωνία για να κινηθούν τα κράτη-μέλη προς την κατεύθυνση αυτή. Και δεν νομίζω ότι οποιαδήποτε μονομερής κίνηση από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είχε πιθανότητες να ευοδοθεί. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Ράντζελ θέλει να κάνει ένα σχόλιο. Κοιτάξτε, θα πρέπει να μιλήσουν και οι συγητέ. Έχει στέχη γιατί πάμε καλά από χρόνο. Θέλω μόνο να πω κάτι σύντομα γιατί μπορεί να δημιουργήθηκε εντύπωση ότι, ε, ότι θέλω να κάνω επανάσταση. Όχι, αυτό που προσπάθησα να εξηγήσω είναι ότι δεν θα πρέπει να βλέπουμε το Κοινοβούλιο σε ένα θεσμό όπου έχουμε μόνο τεχνικούς κανόνες ε, και διαδικαστικούς κανόνες και ότι δεν υπάρχει μια δυναμική μεταλλασσόμενη συνταγματική διαδικασία που είναι διαρκώς εξέλιξη. Ιδιαίτερα να εξετάσει κανείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δει ότι πολλές αρμοδιότητες στην ουσία κατακτήθηκαν από το Κοινοβούλιο και ενώ δεν υπήρχαν πραγματικά στις συνθήκες και αυτό συμβαίνει με κάθε θητεία. Όπως διδάσκω και στους ε, φοιτητές μου, τι συμβαίνει, όπως για παράδειγμα το, ο θεσμός ε, του impeachment ε, στο Αγγλικό Κοινοβούλιο όπου η κυβέρνησή σας ξεκίνησε με αυτή τη νομική διαδικασία που δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική αλλά έχει γίνει πολιτικής φύσης και οδηγεί σε προτάσεις μορφής. Ε, αυτός ο μηχανισμός λοιπόν η λειτουργεί και εδώ και αυτό σημαίνει πιθανότατα ότι σχέσει ανάμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα δεν είναι μόνο νομικής φύσης και αυτό είναι κάτι που ακόμα και το δικαστήριο θα πρέπει να έχει υπόψη του διότι ο θεσμός που είναι πιο δημιουργικό είναι το δικαστήριο και θα πρέπει γι' αυτό το λόγο να καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά τι είναι αυτός ο μηχανισμός. Με αυτή τη λογική την πολιτική και όχι την νομική που προσπάθησε να ε, να πιστήσω την προσοχή σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ σύντομα, τελευταίο σχόλιο. Ναι, σύντομα να πω για το θέμα της λογοδοσίας και της δημοκρατίας και της κοινή γνώμης. Μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε είναι, ε, ε, αυτό μάλλον που προσπαθούμε είναι να κινητοποιήσουμε τον κόσμο εντό του κοινοβουλίου. Δεν ξέρουμε όμω ποια είναι η κοινή γνώμη, γιατί ακόμα και αν το κοινοβούλιο δαπανά εκατομμύρια ετησίω μέχρι το. Ε, με διάφορα μέσα, ποτέ δεν έχει ρωτήσει για το θέμα αυτό. Και έχουμε κάνει έρευνες και λέμε όχι, αυτό είναι ένα θέμα που δεν μπορούμε να το ρωτήσουμε γιατί είναι μέσα στις συνθήκες. Εγώ το θεωρώ τελείω παράλογο αυτό. Ελπίζω να θα καλέσουμε λοιπόν τους εισηγητές να, να βάλουν σε αυτό το την έκθεση το ευρω... και να ζητήσουν αυτό το ευρωβαρόμετρο ότι θα πρέπει να ρωτήσουν τη γνώμη των 25.000 ανθρώπων που ούτω ή άλλω ρωτούν για τις διάφορες στατιστικές τους τη γνώμη τους για την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Εάν δεν έχει κανείς άλλο σχόλιο, από τους ομιλητέ έχετε κάποιο σχόλιο ακόμα να κάνετε. Ναι, για το σχόλιο του κυρίου Ρανζέλ. Ναι, βεβαίως το Ευρωκοινοβούλιο έχει χρησιμοποιήσει τις δημοσιονομικές του εξουσίες για να επεκτείνει τις αρμοδιότητες του στις σχέσεις τις θεσμικές, τις διοργανικές και έχει μεγάλη επιτυχία σε αυτό. ναι, εδώ όμως μιλάμε για ένα τομέα νομοθεσίας όπου μέχρι στιγμή είναι πολύ συγκεκριμένο. Αν δούμε δηλαδή το πρωτόκολλο 6, είναι πολύ ξεκάθαρο το τι περιλαμβάνει και το 10 έχει επίση εκφραστεί. Νομίζω πως το δικαστήριο όταν διαβάζει τη, κανεί την απόφαση του, του 2012 άφησε ανοιχτά διάπλατες τις πόρτες για να αντιμετωπίσει κάποια από τα θέματα. Και αυτό πάντοτε ήταν και η ικανότητα του Κοινοβουλίου να δουλεύει με τις αρμοδιότητες που έχει και κάπως να σπρώχνει, να πιέζει για να αποκτά περισσότερες. Και αυτό είναι και τα τελευταία χρόνια που έχει γίνει. Γι' αυτό και έχουν διευρυνθεί οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου κάθε φορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Ήταν πολύ ζωντανή η συζήτηση ε, και τα σχόλια ήταν πολύ σημαντικά από τους συναδέλφους και τώρα θα ζητήσω από τον, ε, τον κύριο Χέφνερ να κάνει τα τελικά του σχόλια ως συνεισηγητής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους σας και τους συναδέλφους και τους αγαπητούς εμπειρογνώμονές μας που μας βοήθησαν πάρα πολύ σήμερα ε, σε αυτή τη συζήτηση που είχαμε για το θέμα του αντικτύπου της έδρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο δικαίωμά του να αυτοοργανώνεται και να ε, οργανώνεται γενικότερα στα πλαίσια των ε, αρμοδιοτήτων και εξουσιών του. Εγώ δεν θέλω να επαναλάβω όσα υπόθηκαν για να συνοψίσω, ούτε απαραίτητο είναι, ούτε θα ήταν ωραίο. Ακούσαμε πολλά ιστορικά επιχειρήματα, συνταγματικά, εμπειρικά, πρακτικά και ευρήματα, όχι μόνο επιχειρήματα που θα μας βοηθήσουν στην έκθεσή μας. Σε τελική ανάλυση όμως, σε μας εναπόκειται να αποφασίσουμε. Και αυτό που βρήκα ενδιαφέρον είναι ότι στο τέλος φτάσαμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ίσως το κρισιμότερο για όλους μας και ένα κεντρικό ερώτημα. Κάποιοι ε, ζήτησαν επανάσταση. Τώρα ο Ράνζελ είπε όχι δεν εννοούσα εγώ επανάσταση. Να είστε βέβαιοι ότι οι συνεισηγητές σας δεν θα προτείνουν να επαναστατήσει το κοινοβούλιο. Αλλά να είστε βέβαιοι επίσης ότι οι εισηγητές σας θα εξετάσουν σε βάθος τους τρόπους που δεδομένου του συνταγματικού πλαισίου, των συνθήκων, ε, των εξουσιών να κάνουμε βήματα για ένα καλύτερο μέλλον για το κοινοβούλιο μας. Αυτό είναι το κομβικό για όλους. Γιατί πάντα έχουμε την υφιστάμενη, την κείμενη νομοθεσία και τα δικαστήρια που δεν θέλω καθόλου να επικρίνω το δικαστήριο, αλλά το δικαστήριο καλείται πάντα να ερμηνεύει την κείμενη νομοθεσία και οι προγνώμονες βάση αυτής αποφαίνονται. Αλλά ε, σε εμά εναπόκειται να διαμορφώσουμε το μέλλον και ένα κοινοβούλιο που δεν θα εξέταζε σε βάθος τις συνθήκες εργασίας και δεν θα καλούσε βελτίωση, θα ήταν και κακό κοινοβούλιο σε τελική ανάλυση. Θα πρέπει να δούμε πώς επηρεάζει τις ειδικές εργασίες μας αυτή η κατάσταση και χαίρομαι που η ε, ακρόαση αυτή δεν ήταν μεροληπτική, δεν ήταν μονομερής. Ακούσαμε διάφορα επιχειρήματα. Ας πούμε και ένα επιχείρημα που έλεγε ότι αυτό το, το μηνιαίο ταξίδι στο Στρασβούργο είναι ένα είδο ε, κονκλαβίου που επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να οργανωθεί και να ε, συνεδριάσει γιατί δεν υφίσταται την πίεση των ΜΚΟ, των ε, ομάδων πίεσης ή δεν μετακινείται όλο το προσωπικό. Ακούσαμε και άλλα επιχειρήματα και τελικά το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας θα αποφανθεί. Το ξέρω ότι είναι πολιτικό το ζήτημα, αλλά να πω επίσης ξεκάθαρα ότι τις ξέρουμε τις συνθήκες. Έχει αποφανθεί το δικαστήριο μας, έχει εξηγήσει τις συνθήκες και μας είπε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο χειρισμών εντός των συνθήκων. Αν θέλετε λοιπόν χειρισμούς θα πρέπει να αλλάξετε τις συνθήκες. Και θα πρέπει να διερευνήσουμε αν θέλει το Κοινοβούλιο να ζητήσει θεώρηση των συνθήκων, αν ναι, τι είδους. Ακούσαμε διάφορα επιχειρήματα για το τι θα πρέπει να έχετε το δικαίωμα να αποφασίζει το κοινοβούλιο μόνο του και στεναρά επιχειρήματα που λέγουν ότι θα πρέπει να είναι ένα στοιχείο ειλικρινού συνεργασίας. Όλα αυτά θα συζητηθούν, θα συνυπολογιστούν, θα αρχίσει αύριο η συζήτηση και θα συνεχίσουμε ε, βάσει του πρώτου σχεδίου έκθεσης τον Ιούνιο για να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια το φθινόπωρο. Και μου επιτρέπετε να κάνω ένα γενικό τελικό σχόλιο, δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα που πρέπει να τεθεί, υπάρχουν και άλλα πολλά, όπου οι υφιστάμενες συνθήκες δεν πληρούν απολύτως τις προσδοκίες ούτε των πολιτών ούτε των θεσμικών οργάνων. Για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις ε, σημερινές και μελλοντικές. Χρειάζεται λοιπόν τροποποίηση των συνθήκων και συντακτική συνέλευση μετά τις επόμενες ευρωεκλογέ και είμαι βέβαιος ότι το Κοινοβούλιο θα προβληματιστεί σε μεγάλο βάθος για να δούμε τι θα ζητήσουμε εμείς για αυτό το θέμα για τις μελλοντικές συνθήκες. Είδου τι προετοιμάζουμε αυτό το καιρό με τη δουλειά μας, το μέλλον το ίδιο. Και για μένα είναι πολύ μεγάλη πρόκληση για το Κοινοβούλιο, γνωρίζοντας την ιστορία, την ε, παρούσα κατάσταση, να ε, προετοιμάσουμε το μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, για τη συμμετοχή σας. Θα είμαστε σε επαφή, θα παραμένουμε σε συνεννόηση. Αν έχετε άλλες ερωτήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε Μάλιστα, ε, και εμείς ε, οι ίδιοι να έχουμε, οι σκιώδει ηγητές, οι άλλα μέλη, παρακαλώ να μα επιτρέψετε, κύριοι Πυρογνώμονε, να ανατρέξουμε στην πραγματογνωμοσύνη σα. Ευχαριστώ. Τα υπόλοιπα αύριο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρο. Συγχαρητήρια σε όλου του ε, ομιλητέ, ιδιαίτερα στου Πυρογνώμονε και του σπουδαίου συναδέλφου, καθώ και τη γραμματεία που προετοίμασε αυτή τη συνεδρία. Σε ευχαριστώ πολύ και του διερμηνεί και τους τεχνικούς, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να συνεδριάσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.